Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start, uh, and thank you. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθαν. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 13. Μία υπενθύμηση. Σε 11.30 έχουμε το θέμα της Europol και στις 3 το απόγευμα τον διαρθρωμένο διάλογο με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο σας το επισημαίνω για να το λάβετε υπόψη. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, το θέμα των ψυχοτρόπων ουσιών και την υπαγωγή μιας νέας ψυχοτρόπου ουσίας. Η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Λορέντσο Φοντάνα, επειδή το Συμβούλιο έθεσε μια τρίμηνη προθεσμία. αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα αγγλικά για το θέμα αυτό θα ήθελε ο κύριος Φοντάνα να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της εκθεσής του. Η διορία για τις τροπολογίες είναι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Δεν μας έμενε και πολύ καιρός. να μας παρουσιάσει την έκθεση ο κύριος Φοντάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία σύντομη παρουσίαση για το θέμα μας. Για το MDMB, κίμικα. Black Mamba, το 2016 ε, κάναμε μια κοινή έκθεση της Europol και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ναρκωτικών και ε, Εξαρτήσεων Τοξικομανίας. Ε, μετά από το αίτημα της Κομισιόν και 13 κρατών μελών, το Συμβούλιο ζήτησε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που προκαλείται από, τον, από την κατανάλωση του Black Mamba. Πέρα από τους κινδύνους, ζητήθηκε μια μελέτη το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακούν διάφορες οργανώσεις ή μάλλον τι γίνεται με τις εγκληματικές οργανώσεις και τι μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε για τον έλεγχο αυτών των ουσιών. Η Επιστημονική Επιτροπή της OIDT ε, αξιολόγησε τους κινδύνους και στις 28 Ιουλίου του 2016 ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής παρουσίασε στην ε, Επιτροπή και στο Συμβούλιο την αξιολόγηση των κινδύνων και τα βασικά αποτελέσματα είναι ότι αυτό το Black Mamba κατηγοριοποιείται ως ε, συνθετική ανταγωνιστική ουσία των καναβινοειδών είναι γνωστό, γνωστές αυτές ουσίες και ως συνθετικά ε, Από τον Αύγουστο 2014 εμφανίστηκε στην αγορά και εμφανίστηκε σε τουλάχιστον 23 κράτη-μέλη αυτές οι ουσίες. Είναι πολύ ισχυρή αυτή η ουσία. Και έχει ψυχοτρόπες ιδιότητες. Ε, δημιουργεί τεράστιο οξία οξείας ε, τοξικότητας. Οχτώ κράτη-μέλη μίλησαν για 28 θανάτους και 25 περιπτώσεις ε, Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταγραφούν, να καταγραφούν αυτές τις δύο ουσίες στα Μητρώα Ελέγχου των Κρατών Μελών. Ψάξαμε λιγάκι στο ίντερνετ σε ό,τι αφορά αυτές τις ουσίες, αυτή την ουσία και πρέπει να σας πω ότι αυτά που βρίσκουμε είναι σοκαριστικά στο ίντερνετ. Οι συνέπειες αυτής της ουσίας είναι αδιανόητες. Πέρα από τους θανάτους και σοβαρές δηλητηριάσεις, ε, τα άτομα τα οποία δεν πεθαίνουν, ε, μερικές φορές μπορούν να μείνουν ε, ανάπηροι διαβίου. Εξού και η πολύ έντονη επικίνδυνοτητα αυτής της ουσίας. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Φοντάνα. Θέλει παρακαλώ κανείς το λόγο. Η κυρία Ματσόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντικαθιστώ τον Μίχαου Μπόνι. Ο Μίχαου Μπόνι και οι συνάδελφοι του, αλλά και εγώ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φοντάνα για την εκπόνηση και την παρουσίαση της έκθεσης αυτής, του σχεδίου έκθεσης, σε ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για τη νέα ψυχοτρόπο ουσία MDMB SMICA. Αυτή η ουσία θα υποβληθεί στα μέτρα ελέγχου που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιε ψυχοτρόπε ουσίε. Ο κύριο Φοντάνα μας προτείνει την έγκριση της απόφασης και συμφωνούμε. Αυτή η ουσία έχει αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του MCDDA και μάλιστα εντοπίστηκε δραστική αυτή η ουσία σε 23 κράτη-μέλη και 8 μάλιστα έχουν αναφέρει 28 θανάτους και 25 οξύς δηλητηριάσεις και μάλιστα εξαιτία τη υψηλή τοξικότητα ε, και την ε, κειμενόμενη ε, παρουσία αυτή τη ουσία και τη μεγάλη τοξικότητά τη, οι χρήστε δεν μπορούν να ξέρουν κάθε φορά πόσο, τι, ποσότητα δραστική αυτή τη ουσία περιλαμβάνεται σε ένα προϊόν και έτσι δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέπειε. Θεωρείται επικίνδυνη αυτή η ουσία με βάση την εκτίμηση τη ε, αρμόδια ε, υπηρεσία, οπότε συντρέχουν όλε οι προποθέσει για την επιβολή μέτρων ελέγχου. Γι' αυτό και εγκρίνουμε την απόφαση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να εξάρω την σπουδαιότητα αυτής της έκθεσης και να επενέσω το Συμβούλιο για την απόφαση αυτή που έλαβε να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αυτή την δραστική ουσία σε αυστηρούς ελέγχους. Γιατί αν κάθε κράτος αποφασίσει να ελέγξει ή να μην ελέγξει αυτή την ουσία, μια ουσία που είναι ιδιαίτερα τοξική και κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι προφανές ότι ο κίνδυνος ε, επιδεινώνεται. Γιατί υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας ε, στις ε, διασυνοριακές συναλλαγές εντό της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις ελέγχου ή μη ελέγχου. Και για τους νέους παρατηρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μεγάλος αριθμός νέων καταναλώνει τέτοιου είδους ουσίες. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε έκθεση και τη σχετική ε, νομοθεσία που είναι απαραίτητη, ώστε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς εξαίρεση, να εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβαση αυτών των μέτρων. Γιατί θα πρέπει να κριθεί παράνομη η διανομή τέτοιων ουσιών. Αυτό γίνεται προ το συμφέρον των Ευρωπαίων. Θέλουμε να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου και κυρίω του νέου Ευρωπαίου, που είναι ευάλωτη κατηγορία. Ευχαριστώ τον εισηγητή και του εύχομαι καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ, κυρία Γκραπίνη, ευχαριστούμε και τον κύριο Φοντάνα. Όπω σα είπα, αύριο σε 6 το απόγευμα λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα ψηφίσουμε στι 31 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 14 της ημέρησης διάταξης που προβλέπει την παρουσίαση από την Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της απόφασης του 21 Δεκεμβρίου του Δικαστηρίου σε μια συνεκδίκαση υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την συμβατότητα ενωσιακού και εθνικού δικαίου ε, για θέματα διατήρηση δεδομένων και έκδοση θέσεων και κινήσεων, δεδομένων θέσεων και κινήσεων των χρηστών. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας για να μας παρουσιάσει την απόφαση του δικαστηρίου. Ο κύριος Μορ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω σήμερα τις ε, αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2016 ε, του Τμήματος Μίζωνος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά τη διατήρηση δεδομένων από παρόχους ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επίσης την πρόσβαση των εθνικών ε, αρχών σε αυτά τα δεδομένα. Είχαμε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, ε, προδικαστικές παραπομπές από εθνικά δικαστήρια και οι δύο. Η πρώτη περίπτωση ήταν μια παραπομπή ενός ειδικού δικαστηρίου, η υπόθεση Τέλε 2, και η δεύτερη παραπομπή ήταν η υπόθεση Watson και άλλων από ένα Βρετανικό δικαστήριο είναι διαφορετικέ και αφορούν τι εθνικέ νομοθεσίε, τη Σουηδική και την Βρετανική. Αλλά τα ερωτήματα των προδικαστικών ζητημάτων ήταν παρόμοιε, οπότε το δικαστήριο αποφάσισε να τι συνεκδικάσει και να εκδώσει ενιαία απόφαση. Και οι δύο υποθέσει αφορούν την νομιμότητα των εθνικών νομοθετικών διατάξεων για τη διατήρηση των δεδομένων. Η νομιμότητα τέτοιων εθνικών διατάξεων ε, και συμβατότητά του με το ενωσιακό δίκαιο και ιδιαίτερα τι οδηγίε για την ε, ιδιωτικότητα στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η οδηγία αυτή θα πρέπει να ερμηνευθεί υπό το φω και του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό εξέτασε το δικαστήριο. Πριν αναφερθώ στο, στην δικαστική απόφαση να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν μέρο, δεν υπέβαλε, δεν ήταν διάδικο σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπέβαλε παρατηρήσει. Οπότε θα σα παρουσιάσω απλώ την απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα, ω προ τη παραπομπή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολήθηκε με τρία θέματα. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, κυρίω τι οδηγίε για την ε, ιδιωτικότητα σε ηλεκτρονικέ επικοινωνίε. Το δεύτερο θέμα ήταν κατά πόσο η γενική διατήρηση των δεδομένων επιτρέπεται με βάση το ενωσιακό δίκαιο και το τρίτο ζήτημα ήταν οι προποθέσει πρόσβαση των εθνικών αρχών σε τέτοια δεδομένα. Θα αναφερθώ εντάχει και στα τρία θέματα. Το πρώτο θέμα για το πεδίο εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Εδώ το δικαστήριο εξέτασε ε, προσεκτικά τις ε, διατάξεις τις οδηγίες για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και την ερμήνευση υπό το φως του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατέληξε το συμπέρασμα το πεδίο εφαρμογή οδηγίας αυτής καλύπτει όχι μόνο τη διατήρηση των δεδομένων από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά καλύπτει και την πρόσβαση των εθνικών αρχών στα δεδομένα αυτά. Οπότε από αυτή την άποψη το δικαστήριο προβλέπει ευρύ πεδίο εφαρμογής υιοθετεί διασταλτική ερμηνεία δηλαδή για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, το e-privacy. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, γιατί μερικοί θεώρησαν ότι μόνο το πρώτο τμήμα καλυπτόταν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή μόνο τι υποχρεώσει των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στο θέμα όμω τη εσωτερική αγορά, το ενωσιακό δίκαιο ε, είπαν μερικοί, δεν ε, ισχύει για τι εθνικέ αρχέ και κυρίω για την αστυνομία, γιατί τέτοια θέματα εκπίπτουν του ενωσιακού δικαίου. Δεν συμφωνεί λοιπόν το δικαστήριο, απορρίπτει αυτή την ερμηνεία και θεωρεί ότι η σχετική οδηγία καλύπτει και τα δύο σκέλη, δηλαδή και την πρόσβαση των εθνικών αρχών στα δεδομένα. Οπότε ε, η οδηγία είπε ότι εφαρμόζει και το χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ενδιαφέρει άμεσα το Συμβούλιο μια και αφορά νομοθεσία που έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορά συγγνώμη άμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο ε, ζήτημα αφορούσε μια ερώτηση του Σουηδικού Δικαστηρίου που ρώτησε αν είναι δυνατόν να ε, υιοθετηθεί εθνική νομοθεσία που που προβλέπει γενική διατήρηση δεδομένων. Όταν ε, το Συνδικό Δικαστήριο μιλάει για γενική διατήρηση δεδομένων, εννοεί διατήρηση όλων των στοιχείων κινήσεως και θέσεως όλων των χρηστών που αφορούν όλα τα μέσα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δηλαδή, τα πάντα. Τα πάντα θα πρέπει να διατηρούνται συνεχώς. Η... Ο πάροχος Τέλε Tele2 Σβέρικε αντέδρασε σε αυτό το μέτρο, αντιτάχθηκε σε αυτή τη γενική διατήρηση όλων των δεδομένων που χειρίζεται. Η Τέλε 2 Σβέρικε θεωρεί ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο ως θέμα αρχής. Το ΔΕΚ ενέκυψε στο σημείο αυτό και δήλωσε ότι η γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων δεν προβλέπεται από το άρθρο 15 της οδηγίας ε, υπό το φως και του χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων και δήλωσε ότι αυτό υπερβαίνει τα όρια του ότι είναι απολύτως απαραίτητο και δεν δικαιολογείται σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οπότε αυτό που λέει το δικαστήριο είναι σε καμία περίπτωση μια γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Άσχετο αν υπάρχουν άλλα ειχέγγια και ασφαλιστικές δικλείδες για να περάσει κάτι τέτοιο. Αυτό είπε ότι το δικαστήριο τέτοια γενική και διάκριτη διατήρηση δεν επιτρέπεται. Δεν είναι συμβατή με το νοσιακό δίκαιο. Επίσης, αυτή δεν ήταν. Το θέμα είναι πώς ερμηνεύονται οι αποφάσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα. Πολλοί διάδικοι είχαν ερμηνεύσει την ομολογία για τα ψηφιακά δικαιώματα ε, με σωστό τρόπο. Δύο ήταν οι λογικές ε, απόψεις. Η μία έλεγε ότι η γενική διατήρηση δεδομένων είναι δυνατή στο μέτρο που υπάρχουν επαρκείς ε, ασφαλιστικές δικλείδες και στην περίπτωση αυτή ο Γενικός Εισαγγελέας αυτό πρότεινε ότι να επιτρέπεται γενική διατήρηση δεδομένων εφόσον όμως προβλέπονται ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Άλλος Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι η πλειοψηφία των διαδίκων είχαν επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτής της θέσης. Μόνο η μειοψηφία και κυρίως ε, η εταιρεία Τελεδίος Βέριγκε της Σουηδίας ε, ήταν υπέρ ε, της θέσης και του κυρίου Βότσον του Βρετανικού, της Βρετανικής υπόθεσης. Και μόνο η μειοψηφία είπε ότι αν έχουμε γενική διατήρηση δεδομένων αδιάκριτη, είναι απαράδεκτη. Άσχετα με το τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν. Και το δικαστήριο απέρριψε τη σύσταση του Γενικού Εισαγγελέως και τη γνώμη της πλειοψηφίας. Και δικαίωσε την Τελεσβέριγκε και είπε ότι και στην περίπτωση του Βρετανικού Δικαστηρίου αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι η γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων απαγορεύεται ή δεν είναι συμπατή με το νοσιακό δίκαιο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της απόφασης. Επίσης, συνέχισε το δικαστήριο στο σκεπτικό του και είπα ότι ακόμη και αν η γενική και διάκριτη διατήρηση δεδομένων είναι απαράδεκτη, στοχευμένη διατήρηση μπορεί να δικαιολογείται. Και εκεί το δικαστήριο δίνει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για το τι εστί στοχευμένη διατήρηση. Λέει ότι θα πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, σε αντικειμενικέ αποδείξει και τεκμήρια. Και λέει ότι στοχευμένη διατήρηση μπορεί να, να περιορίζεται σε γεωγραφικά κριτήρια, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε περιορισμένο κοινό. Αυτό είναι μια νέα έννοια αυτή τη στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων. Ε, δεν υπήρχε και στα προηγουμένω ε, σε τέτοιε δικαστικέ αποφάσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, την πρόσβαση των εθνικών αρχών σε τέτοια δεδομένα. Εδώ το δικαστήριο ξεκινά από την προπόθεση ότι μόνο στοχευμένη διατήρηση δεδομένων είναι αποδεκτή. Απομένει όμω το θέμα κατά πόσο ε, σε αυτά τα δεδομένα έχουν πρόσβαση οι εθνικέ αρχέ. Και πάλι εξέτασε το δικαστήριο την προηγούμενη ομολογία για τα ψηφιακά δικαιώματα και τον κατάλογο προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούν οι εθνικές αρχές για να έχουν πρόσβαση. Επίσης θα πρέπει να γίνεται λογική, ε, ε, μια λογική αίτηση προς διοικητικό δικαστήριο ή προς δικαστή ή προς διοικητική αρχή και ισχύουν αυτές οι αρχές και μάλιστα είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις και θα πρέπει ε, σορευτικά να τηρούνται. Γιατί μερικοί είπαν ότι ε, μπορούν να τηρούνται και διαζευκτικά. Όχι, το δικαστήριο είπε ότι όλα, όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρούνται, γιατί όλες οι προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να έχουν πρόσβαση οι εθνικές αρχές. Πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση και κυρίως ως προς την ανάγκη να υποβληθεί η αίτηση σε ένα δικαστή για να δώσει την άδεια προκειμένου η Εθνική Αρχή να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Και μάλιστα το δικαστήριο πάει ακόμα πιο μακριά και προσθέτει και νέες ε, προϋποθέσεις και όρους που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη νομολογία για, για τα ψηφιακά δικαιώματα και την Ιρλανδία. Λέει ότι η πρόσβαση μπορεί να ε, επιτρέπεται στα σε εθνικές αρχές μόνο για άτομα που ενέχονται σε σοβαρές ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν υπόνοιες για τέτοια διάπραξη σοβαρού ποινικού αδικήματος. Αυτό είναι μια νέα, πρόθεση, νέα πρόταση, μια νέα ε, προϋπόθεση και μάλιστα παραπέμπει σε πρόσβατη νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπόθεση Ζαχάροφ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο που πρόσθεσε το δικαστήριο είναι ότι από τη στιγμή που έχει γίνει διατήρηση των δεδομένων, τότε οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει να κοινοποιούν του ενδιαφερόμενους ε, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θα θέσει σε κίνδυνο την έρευνα. Και φυσικά αυτοί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα Έχουμε πρόσφατη υπόθεση τρέμς για τα ένδικα μέσα για τις προσφυγές. Οπότε αναπτύσσει περαιτέρω την ομολογία του το δικαστήριο και έχουμε νέες προϋποθέσεις. Πάντω το δικαστήριο αυτή τη φορά διευκρινίζει ότι και οι νέες αρχές και οι προηγούμενες προϋποθέσεις θα πρέπει όλες ορευτικά να τηρούνται. Λοιπόν, κατακλείδη. Η σχετική νομολογία είναι πολύ σημαντική και διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για την, ε, για την ιδιωτικότητα στι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε, που την ερμηνεύει υπό το φω του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποκλείει τη γενική και διάκριτη διατήρηση δεδομένων, αλλά επιτρέπει μόνο τη στοχευμένη διατήρηση δεδομένων. Επίση, διευκρινίζει ποιε είναι οι προποθέσει για την πρόσβαση εθνικών αρχών στα δεδομένα αυτά με βάση την ομολογία για τα, γενικά δικαιώμα, για τα ψηφιακά δικαιώματα δηλαδή και προσθέτει και νέες προϋποθέσεις. Και μία ακόμη παρατήρηση πριν ολοκληρώσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι και πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκε σε νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή. Και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Πολύ συχνά και σε προηγούμενη νομολογία, στην υπόθεση για τα ψηφιακά δικαιώματα και την Ιρλανδία, παρέπεμψε στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα στι υποθέσει ε, Ζαχάροφ για τα μέσα παρακολούθηση ε, στην Ρωσία και Σάμπον Βίση για τα μέσα παρακολούθηση στην Ουγγαρία. Δεν είναι κάτι καινούργιο, λοιπόν η παραπομπή του ΔΕΚ σε νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σαφέ ότι οι νομολογίε και των διαδικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου βρίσκονται στην ίδια γραμμή πλεύση. Αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμε διευκρινήσει, κύριε Μουρ, για τα θέματα τη ε, φύλαξη ε, δεδομένων και τη αδιάκριτη φύλαξη δεδομένων. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι ευρωβουλευτέ ε, έχουν άποψη Προφανώς ε, όλα αυτά που μας είπατε είναι πολύ ξεκάθαρα. Οι βουλευτές ε, θέλουν να δώσουν κάποιες αποχρώσεις σε όλα όσα ακούστηκαν. Νομίζω ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νομική αυτή, αυτή διευκρίνηση και είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ε, ακύρωσε την ε, ε, φύλαξη των δεδομένων, υπήρξε ένα νομικό κενό ή τουλάχιστον νομική αβεβαιότητα και μάλιστα και κατακαιρματισμός. Κάθε κράτος μέλος ανακαλεί την εθνική νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί με βάση την οδηγία για τη φύλαξη των δεδομένων ή όπως έκανε η Σουηδία αξιολογεί ότι η εθνική νομοθεσία ήταν συμβατή με την απόφαση του δικαστηρίου. Αν κατάλαβα καλά τόσα είπε ο κ. Μόρ. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα, γιατί το δικαστήριο είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει γενική υποχρέωση στις ε, εταιρείε τηλεπικοινωνιών να φυλάσσουν δεδομένα διακρίτως. Ε, τι κάνουν όμως τα κρατημέλη τότε, ό,τι θέλουν. Αυτή η περίπτωση με την Τελετούρ και η άλλη υπόθεση του, της, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μήνυμα, είναι σημάδι ότι οι υποθέσεις πλέον θα λύνονται στα δικαστήρια ε, για να εξασφαλίσουμε έτσι ασφάλεια δικαίου και δεν θα την εξασφαλίζει αυτήν την ασφάλεια δικαίου η νομοθεσία. Και αυτό είναι πρόβλημα και για το εθνικό επίπεδο και για την ανταλλαγή πληροφοριών σε τόσο σημαντικά θέματα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου και τις ασφαλιστικές δικλείδες και την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, αλλά είναι και, η ώρα η Κομισιόν να παρουσιάσει μια νέα πρόταση. Είναι επίγον μάλιστα, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε το σοβαρό έγκλημα ή ε, τις απειλές στην δημόσια ασφάλεια, όπως είπε το δικαστήριο, ούτως ώστε να έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα στην Ευρώπη για τη φύλαξη των δεδομένων και να μην ε, παρατηρούμε αυτή την, αυτόν τον κατακαιρματισμό που παρατηρούμε σήμερα. Ευχαριστώ. Κυρία Ζήπολτ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Πάντα ήταν μπερδεμένη η κατάσταση. Μετά την απόφαση για την φύλαξη των δεδομένων, βλέπουμε ότι ο νόμος δεν ισχύει πια, αλλά και οι εθνικές νομοθεσίες, ακόμα και αυτές οι εθνικές νομοθεσίες που δημιουργήθηκαν ως απόρρια της, εθνικ... της κοινοτικής νομοθεσίας, εξακολουθούν να υπάρχουν. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα παραθυράκι, όχι μόνο στο θέμα της φύλαξης των δεδομένων, αλλά και σε άλλους τομείς, όπου έχουμε σύγκρουση με ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν όμω τι καταργήσουμε, τότε μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εθνικές νομοθεσίε. Επομένως, είναι ασαφέ το ποια είναι η νομική βάση, το τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου. Μου άρεσε αυτή η ενημέρωση επίσης, κυρίω σε ό,τι αφορά τις υπερβολές των διοκτικών αρχών. Αυτή τη στιγμή ε, και κυρίως και την πρόσβαση των διοκτικών αρχών. Τώρα δημιουργούμε αυτές τις ε, βάσει δεδομένων και λέμε «Α, οι διοκτικές αρχέ έχουν πρόσβαση σε όλε αυτέ τι βάσει δεδομένων». Μιλάμε για αντιελειτουργικότητα αυτών των βάσεων δεδομένων και αυτή η απόφαση υπογραμμίζει αυτό που είναι τμήμα της συζήτησης ε, στην ομάδα εργασίας ε, για την Αντιελειτουργικότητα και που συζητιέται έντονα ότι χρειαζόμαστε σαφέστατους κανόνες για το ποιος θα έχει πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων και γιατί διάφορες αρχές έχουν πρόσβαση εδώ και εκεί, ας πούμε. Και αυτό ακριβώς υπογραμμίζει την ανάγκη για ξεκάθαρους κανόνες σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ, η Κορνίλια. Η Κορνίλια και μετά η Σόφη. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη διευκρίνηση, παρότι ήταν προφανής η κατάσταση. Η οδηγή ήταν ξεκάθαρη ότι... και έλεγε ότι αν δεν ισχύει πια, δεν ισχύει. Τελεία. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί να ερμηνευτεί. Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα μία απόφαση παραπάνω παρά μία που να μας λείπει και να έχουμε πρόβλημα. Χαίρομαι για αυτή την ε, διευκρίνηση. Και καλό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση για τη φύλαξη των δεδομένων. Όλα όσα αναφέρατε, τα θυμάμαι ότι τα είχα βάλει σε τροπολογίες. Είπα ότι κάποια στοχευμένη φύλαξη είναι αναγκαία όταν υπάρχει υποψία κτλ. κτλ. για κάποιες αξιόπινες πράξεις. Δεν μας αρέσει η στοχευμένη φύλαξη, αλλά το καταλαβαίνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως γενική φύλαξη, γενικευμένη και καθολική φύλαξη. Ακόμα καλύτερα, οι εθνικές αρχές αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Είναι προφανώς λογικό να ξέρουμε τι, θα, τι μπορούν να κάνουν οι εθνικές αρχές. Επιπλέον υπάρχουν και αλυσιδωτές αντιδράσει σε, σε άλλους τομείς, όπως το PNR α πούμε, γιατί αυτό συνδέεται με τη φύλαξη. Μπορείτε να μα πείτε και ποιε θα είναι οι επιπτώσει αν υπάρχουν στο PNR. Και επίση καλό θα ήταν η Κομισιόν να μα πει τι θα γίνει στο μέλλον, εάν οι εθνικέ αρχέ συνεχίσουν χαλαρά, Όπω συνέβαινε μέχρι τώρα α πούμε. Ε, αν έχουμε αυτή την κατάσταση στο εθνικό επίπεδο και αυτή την κατάσταση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τι γίνεται. Φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτά τα θέματα. Είναι τεράστια θέματα. Μην ξεχνάμε ότι η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Και ελπίζω ότι αισθάνονται, αισθάνεται η Κομισιόν πως έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ στην αδελφή. Υπάρχει λογική ε, στο, στην κίνηση της Κομισιόν η οποία έκανε αυτή την ε, πρόταση. Σήμερα το απόγευμα έχουμε και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Ε, φυσικά άλλε είναι οι ερωτήσει του, τη αρμοδιότητά του, αλλά θα μπορούσαμε ίσω να το ρωτήσουμε κάποια πράγματα ε, πέρα από τα δικά του θέματα. Ούτω ή άλλω, ε, ζητάμε, του κάνουμε και διάφορε άλλε ερωτήσει. Θα μπορούσαμε και αυτήν να του την υποβάλουμε. Ε, θα, θα υποβάλω και στον κύριο Μούρ την ερώτησή σα, θα απαντήσει μετά, αλλά η Σόφη τώρα. Ευχαριστώ την νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ κύριε Μουρ για την πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Διάβασα την απόφαση. Ε, τα Χριστούγεννα, θαυμάσιο ανάγνωσμα ήταν. Ενθουσιάστηκα για διάφορους λόγους. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, υπάρχουν διάφορες ε, εθνικές αποφάσεις. Κάποια κράτη-μέλη προσέφηκαν στα δικαστήρια και δέχτηκαν τις ε, συνέπειες. Όχι όλα τα κράτη-μέλη, αλλά σίγουρα κάποια κράτη-μέλη τις αποδέχτηκαν. Δεν είναι μόνο αυτή η απόφαση που έχουμε. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι οι εθνικές νομοθεσίες οι οποίες δεν έχουν, δεν έχουν ανακληθεί μετά την ακύρωση της οδηγίας παραβαίνουν το ενωσιακό δίκαιο. Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τη δυνατότητα μιας νέας πρότασης για μια νέα οδηγία για τη φύλαξη των δεδομένων, αλλά και να εξετάσουμε το δεχόμενο διαδικασία επί παραβάση. Ε, η Κομισιόν έχει και καθήκον για κάτι τέτοιο. Δεν είναι στη εκδητική της ευχαίρεια να αποφασίσει εάν τα κράτη-μέλη ή όχι. Α, χαλαρά μπορούν να παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Κομισιόν πρέπει να παρεμβαίνει. Έχω και ένα πικρό αίσθημα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά όταν η οδηγία πέρασε από το Κοινοβούλιο, εγώ δεν ήμουν από εκείνου που την υποστήριξαν. Δυστυχώ, πολλά από τα επιχειρήματα που είχαμε πει, τότε συμπίπτουν με τα επιχειρήματα του δικαστηρίου στην απόφαση. Η χρήση προσωπικών δεδομένων για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του εγκλήματος, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι αναλογική, στοχευμένη, αναγκαία γιατί θέλετε να ξεπεράσετε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει να δικαιολογείτε αυτό. Αυτό που κάνουν ε, τα δικαστήρια και πολλοί τους ε, κατακρίνουν, τα κατακρίνουν τα δικαστήρια, βασικά είναι να διορθώνουν την κακή νομοθετική μας λειτουργία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε νομοθεσίες που πρέπει να ανακληθούν μετά, θα πρέπει να τις φτιάχνουμε σωστά. Επίσης, τι επίπτωση θα ήθελα να ξέρω θα μπορούσε να έχει αυτή η ιστορία σε άλλα νομοθετήματα και σε διεθνείς συμφωνίε επίσης. Γιατί μπορεί να έχει τεράστιε επιπτώσει, φοβάμαι. Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν η νομική υπηρεσία να χαρτογραφήσει λιγάκι την κατάσταση και τις πιθανές συνέπειες, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες και νομοθετήματα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτή την ιστορία. Τέλο, για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα του δικαστηρίου ήταν η εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η επιχειρηματολογία για να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Καλό θα ήταν λοιπόν να, να κοιτάξουμε τις συνέπειες αυτού του συγκεκριμένου συμπεράσματος σε άλλες πιθανές καταστάσεις. Ευχαριστώ Σόφη. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι προβουλευτές που θέλουν να μιλήσουν, η Ελέν Μίλλερ θα ήθελα να πάρει το λόγο για να απαντήσει ε, και να εκφράσει την άποψη της Κομισιόν και συνεχεί ο κύριος Μουρ για να φτάσει συμπεράσματα. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα και το αίτημα της για την Κομισιόν να αναλάβει δράση. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, να δεσμευτώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση φυσικά αυτή, όπως όλοι ξέρουμε. Και είμαστε σε φάση εξέτασής της. Την αναλύουμε, προβληματιζόμαστε, έχουμε και συζητήσεις και με τα κρατη παράλληλα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, ο Επίτροπος θα έρθει εδώ το απόγευμα, επομένως, αν θέλετε να, έχετε και κάποια πολιτική κατεύθυνση, καλό θα ήταν να υποβάλλετε το ερώτημα αυτό στον Επίτροπο. Φυσικά, αυτά τα σχόλια τα παίρνουμε πολύ σοβαρά και σας διαβεβαιώνω ότι η Κομισιόν θα κάνει το καθήκον της. Όμως δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πολύ πιο λεπτομέρειες και συγκεκριμένη γιατί κοιτάμε τις επιπτώσεις, ευρύτατες ε, επιπτώσεις αυτής της απόφασης σε πολλαπλά μέτωπα. Ευχαριστώ. Δίκιο έχετε. Θα πρέπει να χαράξει μια πολιτική πορεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Σοφή σωστά επισήμενε το καθήκον που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαδικασίες επί παραβάση και τι γίνεται σε περίπτωση που εθνικές νομοθετικές διατάξεις παραβιάζουν ενωσιακό δίκαιο και θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτή τη θέση. Και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Επίτροπο ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μουρ, παρακαλώ, μπορείτε να αντλήσατε κάποια συμπεράσματα και να απαντήσετε και στην ερώτηση Σοφή. Είπε κάποιο πρέπει να ρωτήσει. Ποιον? Εμεί. Εμεί θα ρωτήσουμε. Είπε κάποιο θα πρέπει να ρωτήσει ε, Ναι. Εννοώ, εννοώ. Εμεί. Φυσικά, φυσικά θα ρωτήσουμε. Προσπαθείς πάση θυσία να μιλήσεις έστω και μισό λεπτό επιπλέον Παρακαλώ, σχολιάστε αυτά που ακούσατε για το PNR και άλλες ε, αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά και πώς θα επηρεάσει τη μελλοντική νομολογία ή οτιδήποτε άλλα συμπεράσματα θέλετε να αντιλήσετε μετά τη συζήτηση. Όπως είπαμε, η δικαστική αυτή απόφαση είναι σαφέστατη και ξέρουμε πώς ε, ερμηνεύουμε και την προηγούμενη νομολογία για τα ψηφιακά δικαιώματα και την υπόθεση αυτή με την Ιλανδία. Επίσης, ε, πώς ερμηνεύεται το πεδίο εφαρμογή οδηγίας για την ιδιωτική σφαίρα, ιδιωτική ζωή στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το θέμα της διατήρησης φύλαξης δεδομένων. Δεν εφαρμόζεται μόνο στα σε αυτό το θέμα της διατήρησης δεδομένων, αλλά και σε άλλες υποθέσεις. Ε, ε, θα είναι σημαντική η νομολογία αυτή και σε άλλα θέματα, και όχι μόνο σε αυτό το στενό θέμα της διατήρησης των δεδομένων. Το δικαστήριο μίλησε και εξέτασε πολύ ε, διεξοδικά τις όλες τις διατάξεις ε, για τη διατήρηση των δεδομένων και τη σχετική οδηγία του 2002 και όταν ε, εξετάσαμε την προηγούμενη νομολογία ψηφιακά δικαιώματα Ιρλανδία το είπαμε και το θέμα είναι ότι εφαρμόζεται και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς κανείς μπορεί να αναλύσει σωστά θέματα υπό το φως του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και μας δίνει πολύ ξεκάθαρες γραμμές στο δικαστήριο με την τελευταία του δικαστική απόφαση και θα είναι και πολύ χρήσιμο μοντέλο στο μέλλον που θα το εφαρμόζουμε. Μπορεί να μην καταλήγουμε πάντα σε τέτοια συμπεράσματα. Πάντως το δικαστήριο επιμένει ότι εναπόκειται τώρα στα εθνικά δικαστήρια να εφαρμόσουν και να ε, αξιολογήσουν την εθνική νομοθεσία. Πάντως οι κατευθυντήρε γραμμέ είναι πια ξεκάθαρε. Μπορούμε αυτού του κανόνε να του ε, εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς, το PNR για παράδειγμα, και θα ισχύει και στο, η και για το ενωσιακό δίκαιο και για τις διεθνείς συμφωνίες. Ουσιαστικά αυτό που χρειαζόμαστε μόνο είναι μια επιπλέον δικαστική απόφαση για να δούμε πώς θα εφαρμόζεται και σε άλλου τομεί. Και μάλιστα πολύ φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε τέτοια απόφαση στην υπόθεση Καναδά και PNR. Δεν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί, πάντως αναμένεται όσον ούπο. Και μάλιστα ε, μία εβδομάδα πριν να γίνει η ακροματική διαδικασία για την απόφαση αυτή έγινε για την υπόθεση του Καναδά ε, και ο εισηγητής είναι ο ίδιος. Και μάλιστα επειδή εκ παραλίλου ασχολείται με τα δύο θέματα σίγουρα θα έχει ευθυγραμμισμένη νομολογία. Πάντως πιο γρήγορα ε, διεκπαιρέωσε το προδικαστικό ζήτημα του Σουηδικού και του Βρετανικού Δικαστηρίου. Πάντως στο μέλλον θα έχουμε κατευθυντήρες γραμμές και για την επέκταση σε άλλους τομείς. Και Κάθε δικαστική απόφαση θα την εξετάζουμε φυσικά ξεχωριστά, καταρχήν. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε κάποια συνέχεια αργότερα στις 3 όταν θα έχουμε το διαφορετικό διάλογο με τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 15 για το άσυλο. Η Σιλβίκη Γιώμη είναι εδώ η συγγήτρια. Πρόκειται για την εκπόνηση ενός κοινού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής για τους σκοπού κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος Διεθνού προστασίας. Έχουμε και το σχετικό, τη σχετική νομοθετική πρόταση για την σύσταση του τέτοιου καταλόγου. Στις 26 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Γραφείο Υποστήριξη Ασύλου μία εμπειρογνωμοσύνη για την Τουρκία και στις ε, 16 Νοεμβρίου είχαμε τη δημοσίευση του σχετικού, της σχετικής έκθεσης για την Τουρκία και το καθορισμό του, του καταλόγου ασφαλών χωρών και τα κριτήρια που διέπουν το χαρακτηρισμό της ασφαλούς χώρας καταγωγής. Επίσης, ε, είχαμε την έκδοση ε, έξι εκθέσεων σχετικών για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τώρα θα μας παρουσιάσει ο εκπρόσωπος της του ΕΑΣΟ, του Γραφείου Υποστήριξης Ασύλου, ε, τις σχετικέ εκθέσεις για την Τουρκία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για μια στατιστική επισκόπηση ουσιαστικά αυτών των χωρών και μετά την παρουσίαση της, του ΕΑΣΟ θα γίνει κάποια συζήτηση και θα ακούσουμε φυσικά και την εισηγήτρια την κυρία Κιγιόμ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, thank you um, Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Λούτεν και είμαι ο τμήματάρχης ε, του Γραφείου Ανάλυσης, ε, του Τμήματος Ανάλυσης ε, του ΕΑΣΟ. Δυστυχώς ο διευθυντής του ΕΑΣΟ κολλείεται και τον αντικαθιστώ εγώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε αυτές τις 7 εκθέσεις που, όπως είπατε, δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 και αφορούν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Στην παρουσίασή μου θα σας κάνω μια ιστορική επισκόπηση ως προς το περιεχόμενο για το πώς συντάξαμε την έκθεση, μεθοδολογία, κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης και επίσης θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τις εκθέσεις για κάποια οριζόντια θέματα. Ως προς το, περιεχό, ως προς το πλαίσιο, όπως ξέρετε, σε 9 Σεπτεμβρίου του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για ένα κανονισμό που θα καταρτίζει ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών προέλευσης ε, που περιλαμβάνει όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 λάβαμε και το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χορήγηση εμπειρογνωμοσύνης ως προς την Τουρκία. Και την 1η Απριλίου του 2016 και το Συμβούλιο μας ζήτησε παρόμοια εμπειρογνωμοσύνη και για την Τουρκία και για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το ΕΑΣΟ το γραφείο εμ, να εκπονήσει εκθέσεις ε, για πληροφορίες χωρών προέλευσης για όλες τις 7 ε, χώρες ε, για να γίνει μια στατιστική επισκόπηση των ετούντων προστασία από τις χώρες Νοτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη. Η έκθεση αυτή στηρίζεται σε προσωρινά στοιχεία και με βάση τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και είναι ε, πολύ περιορισμένη η διανομή αυτών των δεδομένων, αλλά έγινα γνωστά στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Περιλαμβάνουμε κάποια βασικά πορίσματα και γραφικές απεικονίσεις ε, το ε, αιτήσεων ε, ασύλου. Και μάλιστα σε, από πρωτοβάθμιες αποφάσεις η περίοδος αναφορά ήταν ε, από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και αφορούν εκθέσεις για τις πληροφορίες χώρας προέλευσης. Οι επτά εκθέσει ε, για τι πληροφορίε χώρα προέλευσης αφορούν την μεθοδολογία που υιοθετούμε για τέτοιε περιπτώσει και περιλαμβάνουν πληροφορίε που συγκεντρώνουμε από ένα ευρύ φάσμα πηγών, και είναι πλήρω εμπεριστατωμένε. Οι εκθέσει αυτέ ε, δεν περιλαμβάνουν εκτιμήσει της ε, ΕΑΣΟ ούτε συμπεράσματα πολιτική στόχο Των εκθέσεων αυτών είναι να παράσχουν πληροφορίες για συζητήσεις επιπολιτικής που θα γίνουν από τους νομοθέτες. Και φυσικά θέλουμε να στηρίξουμε ε, τη συγκεκριμένη επεξεργασία τέτοιων υποθέσεων και τέτοιων αιτήσεων. Τώρα, όρια αναφορά. Χρησιμοποιούμε ίδιου όρου αναφορά και για τι 7 εκθέσει με βάση πληροφορίε που λάβαμε από τα κράτη-μέλη μέσω ερωτηματολογίου για τι ε, εθνικέ πρακτικέ χαρακτηρισμού χωρών ασφαλής προέλευσης του 2015 και σε πληροφορίες που έχουμε λάβει από το στρατηγικό δίκτυο για τις πληροφορίες χωρών προέλευσης. Επίσης έχουμε τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ασφαλούς χώρας προέλευσης όπως προβλέπεται στην οδηγία για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Τώρα εδώ βλέπουμε το συσχετισμό μεταξύ τις οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου και των δικών μας όρων αναφοράς. Και έτσι σας εξηγούμε το σκεπτικό των δικών μας όρων αναφοράς. Η οδηγία για την διαδικασία ασύλου θεωρεί ότι μια χώρα θεωρείται ασφαλής χώρα προέλευσης όταν με βάση την νομική κατάσταση, την εφαρμογή δικαίου εντός ενός δημοκρατικού συστήματος και τις γενικές πολιτικές συνθήκες διαπιστώνεται γενικά και η έλλειψη δίωξη με βάση το άρθρο 9 της Οδηγίας 2011 ε, δεν παρατηρούνται ε, βασανιστήρια ή απάνθρωπη εξευτελιστική συμπεριφορά ή τιμωρία και δεν υπάρχει απειλή λόγω διάκριτης βίας ή κατάστασης ε, διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλη σύραξη. Επίσης, αναφέρεται ότι λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων του εύρου τη Προστασία κατά δίωξη ή κακοποίηση ή κακομεταχείρισης. Τώρα, εμείς ε, δίνουμε κάποιες πληροφορίες ως την ε, κρατική διάρθρωση, το κοινωνικό πολιτικό τοπίο, το κράτος δικαίου, την κρατική προστασία, την κατάσταση ασφάλειας και την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από νομική άποψη γενικώ, αλλά και για συγκεκριμένες ομάδες όπως είναι οι μειονότητες, ε, δημοσιογράφοι, ΜΜΕ, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναίκες, παιδιά, ΛΟΑΔΜΑ, θύματα εμπορίου ανθρώπων, εσωτερικά εκτοπιστέντες και επαναπατριστέντες. Ολοκληρώσαμε την εκπόνηση της έκθεσης το Σεπτέμβριο του 2016 και ε, είναι σημαντικό ότι, ότι έλαβε χώρα μετά την έκθεση αυτή. Φυσικά δεν περιλήφθηκε στην έκθεση. Μία εξαίρεση ε, για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 για την πολιτική ε, που εκδόθηκε σε 9 Νοεμβρίου του 2016. Περιλάβαμε τα πορίσματα της έκθεσής μας Τη έκθεση αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση στη δική μας έκθεση. Μετά την προσέγγιση που είχαμε του δικτύου ΕΑΖΟ για τις χώρες, πληροφορίες χωρών προέλευσης και τις συγκεκριμένε ε, πληροφορίες, καταλήξαμε στις εκθέσεις αυτές μετά τις πληροφορίες που λάβαμε και από τα κράτη-μέλη και μετά από εξέταση ομοτήμων. Εδώ βλέπετε την, τον επιμερισμό του έργου, πώς καταμερίσαμε αυτή, αυτή τη, αυτές τις αρμοδιότητες. Ε, Δεδομένη πίεση χρόνου, δεν πρόκειται να σα παρουσιάσω διεξοδικά το περιεχόμενο και των 7 εκθέσεων. Θα σα δώσω κάποιε πληροφορίε ε, για κάποια οριζόντια θέματα που ε, παρατηρούνται είτε σε όλε, είτε σχεδόν σε όλε τι εκθέσει για τι χώρε προέλευση. Καταρχήν, ο κατάλογος αυτό δεν είναι εξαντλητικός. Οι πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης ε, αναφέρονται ενδεικτικά και οι περισσότερες πληροφορίες, για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπω στις εκθέσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, ούτε ε, εκτιμήσεις κάνουμε, ούτε αξιολογήσεις, ούτε συμπεράσματα συνάγουμε. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι, επαναλαμβάνω, εξαντλητική αυτή η επισκόπηση. Τώρα, αυτός είναι ο κατάλογος των οριζόντιων θεμάτων που έχουν αρκετή σημασία στη συζήτηση για το χαρακτηρισμό των χωρών ασφαλούς προέλευσης. Τώρα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες αυτό. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο στην Τουρκία και στα Δυτικά Βαλκάνια, γι' αυτό υπάρχουν ε, εκθέσεις για διαφορετικά επίπεδα πρόοδου λόγω της ενταξιακής προοπτικής ε, και της ε, πολιτικής απελευθέρωσης. Με βάση τους σχολιαστές Γενικά όμως είμαστε σε αρχική φάση σε αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση, ε, έχουμε εκθέσεις για τις εκλογές που γενικά δείχνουν ότι είναι ελεύθερες και δίκαιες, χωρίς νοθεία. Ε, Επίση, ε, έχουμε διαφορετικά επίπεδα πολιτικής σταθερότητας ή αστάθειας. Στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε συγκρούσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Ε, Έχουμε μποϊκοτάρισμα από την αντιπολίτευση της κοινοβουλευτικής εργασίας ή παραδείγματο χάρη στη ΦΥΡΟΜ, είχαμε ένα μεγάλο σκάνδαλο ε, το, το 2015 με παρακολουθήσεις, συνεχεία πολιτική κρίση και πολιτικό και μποϊκοτάρισμα στο Κοινοβούλιο. Τον Ιούλιο του 2016 ε, είχαμε μία ε, συμφωνία για βουλευτικές εκλογές. Επίσης, στο Κοσμοπέδιο είχαμε μποϊκοτάρισμα ε, από τον Οκτώβριο του 2015. Στο Μαυροβούνιο είχαμε αντικυβερνητικέ ε, διαμαρτυρίες από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά και το Μάιο του 2016 ε, είχαμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση για να οργανώσει τις νέες εκλογές το 2016. Και στα πλαίσια των νέων εκλογών ε, ακούστηκαν ισχυρισμοί για απόπειρα πραξικοπήματο καθώς και ε, χακάρισμα διαφόρων ιστοσελίδων κτλ. στην Τουρκία. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016 ε, θεωρήθηκε επίθεση εναντίον της ε, δημοκρατικά ελεγμένης ε, κυβέρνησης και θεσμών και ανησυχίες όμως εκφράστηκαν για την αναλογικότητα της ε, απόκρισης των αρχών και το κράτος έκτακτης ανάγκης που είχε επιπτώσει στο στρατό, στην αστυνομία, στην στη δημο... στους στη δημόσια διοίκηση, ε, ΜΜΕ, ε, δικηγόρους, ε, εκπαίδευση κτλ. Ε, μιλήσαμε, πολλοί μίλησαν για εκαθάριση. Χιλιάδες απολύθηκαν. Ε, άρθηκε η ασυλία μελών του CHP ε, ε, για τις πληροφορίες για διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας. Υπάρχουν α, καταχρήσεις εξουσίας και στις 7 χώρες. Ε, ορισμένες διαδικασί... Ε, χώρες ε, σημείωσαν πρόοδο, άμεσα την νομοθεσία ή ε, δημιούργησαν θεσμούς κατάλληλους, αλλά η έρευνα και η δίωξη, ας πούμε, εγκλημάτων, η αδικημάτων θεωρείται ανεπαρκής. Επίση, υπάρχει κατάχρηση εξουσία ή υπερβολική άσκηση βία και εξουσία από τι διοκτικέ αρχέ σε πολλές χώρες, ε, ειδικά ε, στην προσπάθεια κατάπνιξης των αντικυβερνητικών ε, διαδηλώσεων. Στην περίπτωση της Τουρκία, οι ισχυρισμοί για υπερβολική βία και παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ακουστεί ευρέω μετά το, την απόπειρα πραξικοπήματο και στα πλαίσια των επιχειρήσεων κατά τη ομοκρατία. Υπάρχουν πληροφορίε για την για μηχανισμούς ε, ανεξάρτητης ε, εποπτείας και παρακολούθησης ε, που ενισχύονται. Φυσικά δεν είναι πάντα πολύ αποτελεσματικοί αυτοί οι θεσμοί και αυτοί οι μηχανισμοί. Η ανεξάρτησία της δικαιοσύνης θεωρείται προβληματική σε πολλές, τις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Παράδειγμα, στην ΦΥΡΟΜ ε, αυτό το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έδειξε την ε, πολιτική παρέμβαση που υπάρχει στη δικαιοσύνη. Μετά την, ε, το πραξικόπημα στην Τουρκία, ε, μαζικές απολύσεις ε, δικαστών έχουν καταγγελθεί. τώρα στα θετικά. Έχουν γίνει κάποιες δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία, Σερβία, Κοσφοπέδιο και Μαυροβούνιο. Αλλά συχνά η εφαρμογή είναι αργή και καθυστερή. Επίσης υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στο διορισμό και την αξιολόγηση των δικαστών, καθώς και πολιτική επιρροή, ε, απόπειρα πολιτικής επιρροής στους δικαστές. Ό,τι αφορά την ε, κατάλληλη κατάσταση ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια, ε, γενικά ε, θεωρούνται ασφαλή παρά τις ε, περίπλοκες διμερείς σχέσεις μεταξύ κάποιων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, Κάποιε ε, τοπικές ε, εντάσεις μεταξύ εθνοτικών ομάδων έχουν αναφερθεί, το Μάιο του 2015 ε, έγινε μια σημαντική, ένα σημαντικό πρόβλημα στο Κουμάνοβο, ε, στην Φιρόμ, όπου ο απελευθερωτικός στρατός του Κωσυφοπεδίου ε, ενεπλάκη, ε, καθώς ε, και η σερβική μειονότητα στο Κωσυφοπέδιο είχε προβλήματα. Επίσης, επιστροφή στη Βοσνία-Σεγοβίνη των μαχητών των ξένων μαχητών, ε, τσιχαντιστών κτλ. Επίσης στην Τουρκία ε, υπάρχει επιδείνωση λόγω τριών πραγμάτων. Στην νότιο-ανατολική Τουρκία από την κατάρρευση της κατάβαση του πυρό τον Ιούλιο του 2015 ε, ακούστηκαν εκθέσεις για στρατιωτικέ επιχειρήσεις σε συνδυασμό με συνεχής ε, ε, απαγόρευση, απαγορεύση κυκλοφορίας. Επίσης, φυσικά, ε, το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου του 2016 που σκοτώθηκαν πάνω από 200 άτομα και συνεχεία ε, η κήρυξη της ε, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Η ελευθεροτυπία στα ΜΜΕ, τεράστιο πρόβλημα δυσυχία και στι 7 χώρε λόγω των ε, συμβάντων, έλλειψης διαφάνειας και στη χρηματοδότηση και στην μεροληπτική παρουσία των ειδήσεων. Ε, συχνά έχουμε περιπτώσεις ε, συκοφαντίας, ε, ε, φυσική βία, ε, κράτηση, ε, κλείνουμε εφημερίδες κτλ, δίμευση, κατάσχεση και δίμευση των περιουσιακών στοιχείων κτλ. Και για τους δημοσιογράφους και για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Τουρκία από το, το δεύτερο εξάμεινο του 2015 παρατηρήθηκε αυτό, αλλά και μετά το πραξικόπημα πάρα πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει. Ε, επίσης, περιπτώσεις παρενόχλησης έχουν αφαιρθεί. Στο κοσφοπέδιο ε, Απειλέ εναντίον δημοσιογράφων έχουν καταγγελθεί και στη Σερβία ε, είχαμε περιπτώσει εκφοβισμού και εκστρατείε συκοφάντηση. Στην ΦΥΡΟΜ ε, είχαμε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και υποκλοπές των δημοσιογράφων στον Μαυροβούνιο, ε, επιθέσεις έχουν καταγγελθεί και δεν, έχουν, ε, ε, δεν έχει θεία άπλετο φω σε αυτά τα περιστατικά κατά των δημοσιογράφων. Επίση, εκφοβισμοί στη ε, δημοσιογράφων στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σε ό,τι αφορά τι εθνικέ και θρησκευτικέ μειονότητε, διακρίσει εναντίον των Ρωμάν, των Ασκάλι και των Αθήγκανων έχουν αναφερθεί για όλε τι χώρε των Βαλκαν... Βαλκανίων, πρόσβαση στη στέγη, στην υγεία και στην αγορά εργασία είναι προβληματική. Ε, επίσης, έχουμε ε, Ρωμά ε, σε δύσκολη κατάσταση στην, ε, στο Μαυροβούνιο. Επίσης στην Τουρκία έχουμε διακρίσει εναντίον τους, των Ρωμά και των ΣΥΑ και των Αλεβί. Για τους Κούρδους ε, πρόσφατα ε, έγιναν διάφορες μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσουν τα δικαιώματά τους στην Τουρκία, αλλά όμως μετά την, κατάπαυση της, ε, την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός το 2015 υπάρχουν προβλήματα στην κατάσταση. Η κατάσταση των σεξουαλικών δυνοτήτων είναι τεράστιο θέμα ανησυχία στις περισσότερες χώρες. Έχουν γίνει καταγγελίες για διακρίσεις, ρητορικέ μίσου από εκτρεμιστέ ή ή θηκεφτικέ ομάδε, αλλά και πολιτικέ, ε, πολιτικούς, ε, παρενόχληση από αστυνομία, αλλά και φυσική βία. Η θρησκευτικε ομαδε αλλα και απο πολιτικου πολιτικους ε παρενοχληση απο την αστυνομια αλλα και φυσικη βια η αντιδραση των διοκτικών αρχών κατά των εγκλημάτων των ε, ΛΟΑΔ συχνά θεωρούνται έτσι πολύ χαλαρές, πολύ ήπιες. Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά μέτρα κατά των διακρίσεων. Υπάρχει μεγαλύτερη αφύπνιση ε, στο πληθυσμό. Ε, Παραδείγματο χάρη στο Κοσμοπέδιο. Ε, είχαμε στο Κοσμοπέδιο Μα, Μαυροβούνιο, Αλβανία, ε, πορείες gay pride και τέτοια. Ε, επίσης, το τελευταίο οριζόντιο θέμα αφορά την κατάσταση των παιδιών και των γυναικών. Ε, η, η συζυγική βία, η βία στο σπίτι ε, είναι ανησυχία σε όλες ε, τις χώρες, παρά τα θετικά μέτρα που υπάρχουν σε διάφορες χώρες υπό τη μορφή σχεδίων δράσης, ε, εκστατιών αφύπνισης και της δημιουργίας ε, καταφυγίων για τις γυναίκες. Πολύ γάμοι σε μικρή ηλικία είναι έντονοι στην Τουρκία, αλλά και στους Αθήνκανους των Δυτικών Βαλκανίων εν γέννη. παιδική εργασία είναι ευρεία στην Τουρκία, παρά κάποια θετικά μέτρα. Ε, και σε πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, έχουμε καταγγελίες για ε, καταναγκαστική εργασία για παιδιά Ρωμά. Επίσης, σεξουαλική βία και σωματεμπορία παρά κάποια θετικά μέτρα έχουμε. Παρακαλώ, με αυτά τελειώνω την παρουσίασή μου, αλλά μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση COI και για τις 7 χώρες μεθοδολογία δηλαδή για τις χώρες προέλευσης. Εγώ σας δίνω μία απεικόνηση απλώς ε, ε, και μία σύνοψη όλων αυτών των εκθέσεων που έχουμε για διάφορα θέματα. Ε, σας είπα τη μεθοδολογία. Προσπάθησα να εξηγήσω κάποιες ερωτήσεις για το περιεχόμενο. Δεν θα κάνω καμία όμως αξιολόγηση για την ουσία των, ε, της κατάστασης της χώρας αυτές, γιατί αυτό είναι καθήκον των συνομοθετών. Σας ευχαριστούμε. Όπως είπατε κι εσείς, το πολιτικό καθήκον ε, της εξέτασης ε, της έκθεσης του Άσο ανατίθεται στους, στη και στους α, πολιτικούς, βουλευτές. Κύριε Γκυγιώμη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, οργάνωση αυτής της ε, συζήτησης και θα ήθελα να χαιρετήσω ε, το έργο των επιτελείων του ΕΑΣΟ και για την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών. Δεν φαίνεται από τις διαφάνειες, αλλά είναι πολύ μεστές και άρτιες αυτές οι εκθέσεις και πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε καθημερινά προκειμένου να στηρίξετε τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Πολιτικής Ασύλου. Θα θυμάστε το έργο ε, για το κατάλογο, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο ε, για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης. Συνεχίζονται οι εργασίες, υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιοι σκόπελοι, θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Αλλά, όπως είπατε, πρόκειται για μερική εντολή. Δηλαδή και εμείς και το Συμβούλιο συμφωνήσαμε ως προς τη βασική δομή του καταλόγου. Αυτό είναι το θέμα το τυπικό και το θέμα του περιεχομένου είναι το, θέμα, το δεύτερο θέμα. Και ζητήσαμε μια υπερογνωμοσύνη από το ΕΑΣΟ γιατί θέλουμε μια σοβαρή ανάλυση κατάστασης. Όχι γιατί η αρχική αξιολόγηση της πρότασης δεν ήταν σοβαρή, αλλά θεωρήσαμε ότι τα κριτήρια δεν ήταν αρκετά και δεν ήταν αρκετά εμπεριστατωμένη ανάλυση. Γι' αυτό ζητήσαμε πιο διεξοδική επισκόπηση των προτινόμενων χωρών. Μας δώσατε αρκετές πληροφορίες που δεν ε, ε, ανταποκρίνονται στην πυκνότητα των εκθέσεών σας και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να διαβάσουν ε, ολόκληρες εκθέσεις. Είναι πραγματικά αμερόληπτη παρουσίαση των στοιχείων και πολύ μεστή, επαναλαμβάνω, παρουσίαση και μάλιστα ο κατάλογος αυτός των, χωρών, των ασφαλών χωρών προέλευσης ε, δεν συνοδεύει τις μεταναστευτικές ροές, αλλά καθιστά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χορήγησης Ασύλου πιο αποτελεσματικό. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπατε και οι διαπιστώσεις που κάνατε, η παρουσίαση ε, των στοιχείων που μας κάνατε, δείχνουν ε, οπωσδήποτε την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων και είναι αδιαφυσβήτητο ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα στην Τουρκία ε, με μεγάλη διαφορά μεταξύ Τουρκίας και των υπόλοιπων έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ε, περίτρανη, εμφανέστατη αυτή η διαφορά μεταξύ Τουρκίας και χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και ελπίζω να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι διαφορές για να ολοκληρωθούν ε, οι τριμερείς διάλογοι μετά τη φιλόδοξη στάση ε, που υιοθετήσαμε και υπερψηφίσαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σιλβί, γιατί πραγματικά ε, έθεσε σωστό πλαίσιο αυτή τη συζήτηση για την έκθεση, για τις πληροφορίες, για τις χώρες προέλευσης. Από το ΕΛΚ η κυρία Τατή είναι η σκιώδη συγγήτρια, δεν έχει έρθει ακόμη όμως. Ο κύριος Δεπρέ είναι ο σκιώδης συγγητής από τους φιλελεύθερους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση του τμήματάρχη του ΕΑΣΟ και τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση. Δυστυχώς δεν έχω διαβάσει το σύνολο των εκθέσεων και έτσι δεν μπορώ να αποφαθώ επί της ουσίας. Μετά από την ε, παρουσίαση πάντως ε, διαπίστωσε ότι υπάρχουν κάποια οριζόντια σημεία σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Ε, προβλήματα έχουμε και στις 7 χώρες σε ό,τι αφορά το σεβασμό των μειονοτήτων. Διακρίσεις ε, παρατηρούνται σε όλες τις χώρες επίσης. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τους ΛΟΑΔΜ, ανησυχητική είναι η κατάσταση σχεδόν σε όλες τις χώρες επίσης, τις 7. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών και παιδιών, υπάρχουν φαινόμενα ενδοικογενειακή βίας, ε, βίας κατά των γυναικών. Και αυτό εμφανίζεται σε όλες τις χώρε το φαινόμενο. Τα πρώτα σημεία δεν τα ανέφερα καν. Οπότε η πρώτη μου αντίδραση είναι μένουμε εμβρόντιτοι με τα συμπεράσματα αυτά είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αυτές τις χώρες ως ε, ασφαλείς χώρες ε, προέλευσης. Θα προτιμούσα η ανάλυση που κάνατε εσείς να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν υποβάλει τη σχετική έκθεση. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο συνεπές και πολύ πιο συγκροτημένο από αυτό που έγινε, αυτό το προθύστερο που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι η εντολή είναι μερική. Δηλαδή δεν συζητούμε για τον κατάλογο καθ' αυτό. Οπότε ρωτώ, τι ακριβώς γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, δεν το λέω σε εσά. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνομαι. Γιατί φαντάζομαι ότι θέλουμε κάποια συνέπεια. Έχουμε 7 χώρες που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την ανάλυση της κατάστασης ε, που παρουσιάζει ε, η ΑΣΟ, κανονικά καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει θέση σε κατάλογο ασφαλών χωρών. Και σίγουρα όχι η τελευταία που προσθέθηκε εκ των υστέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα για διευκρίνηση τους λόγους. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι ακριβώς επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση αυτή. Και πραγματικά μπράβο στην εισηγήτριά μας που με ιδιαίτερο ζήλο υπεράσπισε τη θέση τη δική μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ευχαριστώ για την προσήλωσή της σε αυτό το θέμα και την συγχαίρω επευκαιρία και για την επανεκλογή της ε, στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, φαντάζομαι ότι το υψηλό σκορ που είχε εξηγείται από την σύσσωμη υποστήριξη που της έδωσε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είμαι σχεδόν βέβαιο γι' αυτό. Λοιπόν, σε τι σενάριο προσπαθεί να μα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι παίζουμε ακριβώ εδώ. Γιατί ε, πρόκειται για μερική εντολή. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, ε, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο κατάλογος των ασφαλών χωρών. Οπότε τι θα προτείνει ε, στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω ξεκάθαρη παρουσίαση των πραγμάτων. Τι σενάριο παίζεται εδώ. Δεν θέλω να μας κοροϊδεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Ξέρω γιατί συνεχάρη στην κυρία Γεγιόμ, γιατί έχει πολύ ε, συγκεκριμένο έργο και ε, σίγουρα δεν χρειάζεται καν να ακούμε την παρουσίαση της ΕΑΣΟ αρκεί να ανοίξει κανείς την τηλεόραση και βλέπει τι κατάσταση επικρατεί σε αυτές τις χώρες που αποκαλούνται μερικές φορές ασφαλείς χώρες προέλευσης. Και ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τη ΕΑΣΟ που μας έδωσε μια σαφή επισκόπηση της κατάστασης, αλλά γνωρίζουμε όλοι περί τίνο πρόκειται, γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση επικρατεί στι χώρε αυτές. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ποιότητα και η αρτιότητα αυτών των εκθέσεων. Θα πρέπει τώρα να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς όλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στην κυρία Μποντήλ Φεραίρο πριν ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του ΕΑΣΟ για την πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση της κατάστασης και την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των εκθέσεων αυτών. Εγώ δεν ήμουν πολύ αισιόδοξο προ την ίδια την έννοια της ασφαλού χώρας προέλευση. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανεί ότι η Σουηδία είναι ασφαλή χώρα και παρόλα αυτά πολλοί δεν θέλουν να πάνε εκεί. Οπότε πώ μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την έννοια τη ασφαλούς χώρα. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να γίνει μια περιπτωσιολογική ανάλυση της κάθε κατάστασης. Και αυτό είναι ο στόχος. Και συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια του κυρίου Ντεπρέ εδώ έχει γίνει ένα προθύστερο σχήμα. Ανάποδα. Ξεκινάμε από το τέλος. Πρώτα θα έπρεπε να δούμε ε, τις συνέπειες μιας πρότασης και μετά να την υποβάλουμε. Ενώ εδώ πρώτα η πρόταση και μετά να λύουμε τις συνέπειες. Και τελικά, ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να καταργήσουμε αυτό το κατάλογο ασφαλών χωρών και να εξετάζουμε περιπτωσιολογικά κάθε χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο δικαίωμα του καθενός και έτοιμα θεμητό. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών και η Τουρκία σίγουρα είναι από τις λιγότερο ασφαλείς χώρες και παρόλα αυτά υπάρχει στον κατάλογο. Αλλά και οι υπόλοιπε χώρες ε, ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διαφορετικό βαθμό. Οπότε, με βάση αυτήν την έκθεση, τι συμπεράσματα να αντλήσουμε. Τα δικά μου συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να καταργήσουμε όλο χερό αυτόν τον κατάλογο ασφαλών χωρών. Ευχαριστώ. Ρομπέρτα, θες να μιλήσει ξανά ονόματο τη κυρία Ντάτη. Ναι, δεν μπόρεσε να έρθει καιρό, ζητάει συγγνώμη. Θα διαβάσω την παρέμβαση τη στα γαλλικά. Πρόεδρε, συνάδελφοι, σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους α, ομιλητές. Έχει πει πολλές φορές η κυρία Σιλβική Γιώμη και οι σκιώδησίτες το ότι ο ρόλος της ΕΑΖΟ και η μεθοδολογία είναι σημαντική για την σύσταση αυτού του καταλόγου ασφαλών χωρών. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται ε, για κάθε χώρα η οποία μπαίνει σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να είναι ο πιο μακρύ δυνατό αυτό ο κατάλογο, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματική η μεταναστευτική μα πολιτική. Είναι σημαντικό να έχουμε και για τι 7 αυτέ χώρε που προτείνει η Κομισιόν μια αιτιολόγηση. Ε, προτείνεται ότι είναι σίγουρε χώρε. Ζητάμε. Ο, ζητάμε ε, λυπούμαστε όμως που καθυστέρησε πολύ δημοσίευση για, τα, για την έκθεση για την Τουρκία. Εμείς τώρα θα αποφασίσουμε τι συνέχεια θα δώσουμε. Γιατί έχουμε, εδώ υπάρχουν πολιτικά ε, και διπλωματικά διακυβεύματα. Ε, αυτό το ντοσιέ ε, καθυστερεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ μακρές. Ζητώ από τη Μαλτέζικη Προεδρία να δείξει πραγματική βούληση για να επανεκκινήσει τις ε, συζητήσεις για τον καονισμό, δύσκολες συζητήσεις, για να πεμπλακεί το θέμα. Ε, τη στιγμή που η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική εγείρει μείζονες ανησυχίες στους πολίτες μας. Γι' αυτό ακριβώς κανένα δεν μπορεί να ξεχάσει τις ευθύνες του. Όλοι είμαστε αντιμέτωποι με αυτές. Ευχαριστούμε Ρομπέρτα. Πρώτα θέλω να δώσω το λόγο σε κάποιον από την Κομισιόν και συνεχεία θα δώσω το λόγο πίσω στην κυρία Γκυγιόμ για να κλείσει το θέμα αυτό. Υπάρχει άτομο από την Κομισιόν. Καλημέρα. Ακούσα μεγάλο ενδιαφέρον την ε, παρουσίαση του ΕΑΣΟ και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. Σε ό,τι αφορά τη θέση της Κομισιόν, την ξέρετε, εμείς κάναμε την πρότασή μας εδώ και καιρό. Κάναμε τότε και την αξιολόγηση ότι αυτές οι 7 χώρες στον προτινόμενο κατάλογο πληρούν τις α, συνθήκες που αναφέρει η οδηγία για το άσυλο για να θεωρηθούν ασφαλείς. Ο λόγος ε, για τον οποίο θεωρούμε ότι είναι ασφαλείς χώρες ε, αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη της πρότασης. Χαιρόμαστε λοιπόν για την συνεισφορά του ΕΑΖΟ σε όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι μια καλή βάση, ούτως ώστε οι συνομοθέτες με βάση και αυτά τα στοιχεία να συναποφασίσουν. Αλλά τώρα πια το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των συνομοθετών. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. λέει ο πρόεδρο. Δεν φανταζόμασταν ότι με αυτή την παρέμβαση θα λυνόταν όλα τα προβλήματα. Θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στη Σιλβίκη Γιόμ. Δεν αμφισβητούμε καθόλου τις, ε, την ορθότητα των εκθέσεων. Το πρόβλημα ποιο είναι, αυτό που βλέπουμε όλοι και δεν το λέμε. Ότι ξέρουμε την κατάσταση σε αυτές τις χώρες, την πολιτική κατάσταση, Και θα ήθελα να μας πει η Σιλβή Κιγιόν πώς, κατά την άποψή της, πρέπει να προχωρήσουμε. Σύντομα. Σε σχέση με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Με αυτού του συναδέλφους ούτως ή άλλως έχω συζητήσει το θέμα διαμακρών. Και βλέπω ότι επαναλαμβάνω τι θέσει που έχουν ήδη πει. Έστω και αργά, γιατί η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλη, κολοσιαία θα έλεγα, έστω και βλεπω οτι επαναλαμβανω τις θέσει που εχω ηδη πει εστω και αργα γιατι η δουλεια που πρεπει να γινει ειναι παρα πολυ μεγαλη κολοσιαια θα ελεγα εστω και αργα έχει νόημα. Γιατί θα μας βοηθήσει αν προκύψει τέτοιο ευρωπαϊκός κατάλογος ασφαλών χωρών για να ξεκαθαρίσουμε τις ιδέες για το πώς θα συντάξουμε αυτόν τον κατάλογο. Νομίζω ότι ήταν ένα βασικό θέμα των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε το γεγονός ότι δεν λάβαμε υπόψη μας ότι η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και η σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Ασφαλών Τρίτων Χωρών παίζει ένα ρόλο στη μεταναστευτική πολιτική, στη διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ε, κανονικά δεν φτιάχνεται γι' αυτό ένα κατάλογος. Και δυστυχώς ένας από τους βασικούς κοπέλους είναι ότι αυτή η πρόταση έγινε εν μέρη ακριβώς για την μεταναστευτική πολιτική τελικά. Το θέμα του ασύλου και του δικαιώματος ασύλου. Ε, γι' αυτό γίνεται ε, και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Προηγουμένως έμεσα είπα τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το φάκελο. Δεν είμαστε εδώ σήμερα γι' αυτό. Θα επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο θέμα κάποια στιγμή. Αλλά φυσικά έχουμε τρομερά έξοδα. Η θέση της Επιτροπής ε, Λίμπε στο παρελθόν ήταν πολύ στεναρή και φιλόδοξη. Ξεκινήσαμε τις ε, συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου και για τα τέσσερα βασικά κεφάλαια που εντοπίσαμε, δύο, σε δύο από αυτά έχουμε τεράστια προβλήματα μπλοκάρισμα θα έλεγα. Ένα παράδειγμα, υπάρχουν και άλλα. Η ιδέα ότι, μπορούμε, ότι δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε, το λέει το Συμβούλιο, τους εθνικούς καταλόγους, ποτέ δεν τους εγκαταλείπουμε, ακόμα και αν έχουμε τον ε, ευρωπαϊκό κατάλογο, με κοινά κριτήρια και κοινό στόχο Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να μην υπάρχουν πια, εφόσον έχουμε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο ή Εθνική Κατάλογο. Αλλά το Συμβούλιο επιμένει να του διατηρήσει. Επομένω, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια φιλοδοξία και απαιτητικότητα στην έκθεση για τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου. και θα πρέπει να λάβει υπόψη το περιεχόμενο ε, της έκθεσης για το θέμα του καταλόγου ασφαλών τρίτων χωρών. Θα συνεργαστώ με τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές για να δω τελικά τι περιεχόμενο θα λάβει η έκθεση για τις διαδικασίες. Ευχαριστώ Σιλβί. Χρήσιμη η συζήτηση μας έδειξε την προσέγγιση σε αυτόν τον κοινό κατάλογο και η Σιλβή μας είπε ποια είναι η θέση της. Μας μίλησε για τους τριμερείς διαλόγους. Ούτως ή άλλως θα γίνει μια... Έγινε και θα γίνουν και άλλες ε, ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις. Και ούτως ή άλλως οι εκθέσεις αυτές ήταν χρήσιμες παρά την χρονική στιγμή στην οποία υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για τις συνεισφορές τους. Ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Φτάσαμε στις 11 και 7. Το επόμενο σημείο είναι τεράστια τεχνική σημασία για την Επιτροπή μας και πολιτική σημασία και ξεκινάει στις 11.30. Γιατί χρειαζόμαστε τους συναδέλφους από το Συμβούλιο και την Κομισιόν παρόντες. Δεν είναι όμως εδώ ακόμα, γι' αυτό ακριβώς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα ξαναρχίσουμε στις 11.30 Dan. Παρακαλώ να είστε στην ώρα σας για να ξεκινήσουμε το σημείο 16. 11.30 παρακαλώ.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

Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 16. Όπως ξέρετε, είναι ένα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι παρόντες. Ε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κάποιοι από εσά θα γνωρίζουν το ζήτημα, κάποιοι όμως ε, ίσως όχι, οπότε θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή και θα εξηγήσω πού βρισκόμαστε. Θα συζητηθεί και στην ιδρύα των συντονιστών το θέμα αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλήρη και διαφανή συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση εδώ σήμερα στην Επιτροπή μας για να δώσουμε έτσι γραμμέ γραμμές προς την συνάντηση των συντονιστών. Όπως ξέρετε η Δανία δεν θα μπορέσει να συμμετέχει πλέον στη Europol την 1η Μαΐου του 2017 με βάση τον νέο κανονισμό της Europol μετά την αρνητική ε, έκβαση του ψηφίσματο του 2015 στην Δανία, ξεκίνησε διαπραγματεύσει μεταξύ Δανία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι ώστε η Δανία ε, να μπορέσει να είναι όσο γίνεται πιο στενά συνδεδεμένη με το Europol ε, εντό εισαγωγικών. Αυτό κοινή δήλωση 15 Δεκεμβρίου ε, του κ. Γιούγκερ, του κυρίου Τάσκ και του Δανού Πρωθυπουργού είχαμε. Στην κοινή αυτή δήλωση προτάθηκε για να αποφύγουμε ε, τα επιχειρησιακά κενά η σύνδεση της Δανίας με την Europol να πάρει μια μορφή ε, συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ Δανίας και ε, Europol πριν από το Μάιο του 2017. Με βάση λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου για την Europol. Εδώ έχουμε δύο διαδοχικές νομοθετικές διαδικασίες. Θα συζητήσουμε την πρώτη σήμερα. Η Δανία λοιπόν θα μπει σε ένα κατάλογο με τις χώρες με τις οποίες η Europol μπορεί να συνάψει διεθνείς συμφωνίες και στη συνέχεια θα έχουμε τη Συμφωνία Επικρισιακής ε, Συνεργασίας με τη Δανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια ε, θα δώσει τη γνώμη του σε αυτές τις διαδικασίες. Όπως ξέρετε, επιτάπητος εδώ ε, έχουμε μια απόφαση εφαρμογής, εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου που έχει να κάνει με τον πρώην τρίτο πυλώνα, πριν τη Λισαβόνα δηλαδή, πέρα από το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι πολύ σφιχτό, όπως θα ξέρετε θα τεθούν και κάποια πολιτικά και νομικά ζητήματα αρκετά σημαντικά. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να το συζητήσουμε αυτό όσο γίνεται πιο ανοιχτά και να δούμε ποια οδό θα ακολουθήσουμε για να επιληθεί αυτό το πολιτικό και θεσμικό ζήτημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα γίνει παρουσίαση σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την Προεδρία και από τις Δανικές Αρχές. Έχει γίνει μια προπαρασκευή πριν από τη συνεδρίαση αυτή εν ώψη της σημερινής μας ε, συνάντησης είναι σημαντικό πάλι στα μέλη της Επιτροπής μας να πούν σαφώς ποια είναι η θέση τους για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία και στον εκπρόσωπο της δανική Κυβέρνησης. Πρόκειται για έναν ανώτατο αξιωματούχο της ε, δανική Δημόσιας Διοίκησης που θα μας παρουσιάσει τα διάφορα επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν τη χώρα του. Θα έχουμε μια συναντρία των συντονιστών μετά από αυτή τη συνεδρίαση και αυτή τη συνεδρίαση των συντονιστών θα αποφασίσουμε γύρω από μια σειρά από Να το πω όμως από τώρα, για να υπάρχει πλήρη διαφάνεια, θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο συγητής για την γνωμοδότηση. Θα πρέπει επίσης να αποφασίσουμε κατά πόσο έχουμε κάποια νομική ε, γνώμη επί του αυτού και δεν θα πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις. Και βέβαια σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις αρμοδιότητές μας θα πρέπει σε ένα ψήφισμα να λέμε σαφώς ε, να επαναλαμβάνουμε τις αρμοδιότητές μας και να τονίσουμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση ad hoc. Καλό είναι οι συνάδελφοι να γνωρίζουν λοιπόν όλα αυτά τα αισθήματα που θα συζητήσουν οι συντονιστές. Μετά από αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λουίτζι, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και καλημέρα σε όλους όλες, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελευθεριών. Ο Πρόεδρος ήδη ε, έκανε μια εισαγωγή στο ζήτημα. Δεν θα επανέλθω εγώ στο θέμα του πρωτοκόλλου 22 ε, και στο γεγονός βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή σέβεται απολύτως τη δημοκρατική επιλογή του δανεικού λαού του Δεκεμβρίου του 2015. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι από την 1η Μαΐου 2017, όταν δηλαδή ο νέος κανονισμός Europol θα τεθεί σε ισχύ, η Δανία δεν θα αποτελεί πλέον μέλος της Europol. Και θα θεωρείται μια τρίτη χώρα σε σχέση με την Europol. Αυτό σημαίνει ότι η Δανία δεν θα δεσμεύεται από τον κανονισμό Europol και από την 1η Μαΐου δεν θα υπάρχει πλέον ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία με τη Δανία ε, και μεταξύ της Δανίας και της Europol των άλλων 27 κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση λοιπόν ήταν να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, να αντιμετωπίσουμε επιγόντως το θέμα αυτό για το καλό όλων ε, των συμπολιτών μας και των δανών συμπολιτών μας. Δεν θέλω να μπω στην περίπλοκη κατάσταση σε πεδο ασφάλειας ε, που ζούμε σε μια προσπάθεια να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτή η κατάσταση ασφάλειας έχει, ε, έχει νέες διαστάσεις, οπότε είναι ανάγκη υπάρχει ανάγκη όλα τα κράτη-μέλη να είναι ενεργά αλλά και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή τους. Δεν πρέπει λοιπόν η Δανία να γίνει έτσι το αδύναμο σημείο στην συνεργασία στα πλαίσια της Europol. Επίσης πρέπει να αναγνωριστεί ότι η Δανία είναι ένα σημαντικός εταίρος για την ε, εφαρμογή του νόμου. Είναι βασικός ε, συνεισφορέας στην βάση δεδομένων της ε, Europol. Να δώσω κάποια στοιχεία ενημερωτικά. Σε ό,τι αφορά συνεισφορά στη Europol και το σύστημα πληροφοριών της Europol, ανά εκατομμύριο κατοίκων, η Δανία είναι στην 7η θέση μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό βεβαίω είναι αρκετά αξιοσημείωτο. Επίσης, είχε 1.200 συνεισφορές ε, στους φακέλους ανάλυσης της Europol και συμμετείχε σε 25 από τις 29 από 25 από τα 29 σημεία εστίασης της, Κομισιόν, της Europol. Ένας πολύ υψηλός αριθμός. Επίσης, ε, συχνά η Δανία ανταλλάσσει εμπειρογνώμονες και πραγματογνωμοσύνη. Ε, συμμετέχει ενεργά στην πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων. Ο πρόεδρος Γιούγκερ, λοιπόν, από με τον πρόεδρο Τάσκ, και τον Δανό Πρωθυπουργό Ρασμούσεν συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο διακανονισμό, ε, κάποιο επιχειρησιακό διακανονισμό για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τι αρνητικέ επιπτώσει τη ε, αποχώρηση τη Δανή Europol από την 1η Μαου. Θεωρούμε σκόπιμο να δώσουμε τη δυνατότητα συνεργασία μεταξύ Europol και Δανία σε σημεία κλειδιά έτσι ώστε η Ένωση αλλά και η Δανία να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ε, απειλές για την ασφάλειά τους. Στις 15 Δεκεμβρίου η δήλωση προβλέπει ένα διακανονισμό ε, που θα αφορά τη Δανία και μόνο τη Δανία ε, και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν ισοδυναμεί με πλήρη συμμετοχή στην Europol. Θα πρέπει να υπάρξει μια επαρκέ επίπεδο συνεργασία με τι δανεικέ αρχέ επιβολή του νόμου και σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή δεδομένων Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλε δικλείε ασφαλεία. Η συμφωνία πάντω ε, την οποία έχουμε κατά νου δεν πρέπει και δεν μπορεί να δίνει πρόσβαση στι δανεικέ αρχέ ε, στα δεδομένα τη Europol και στα αρχεία τη Europol, ούτε πλήρη συμμετοχή στο επικοινωνιακό έργο τη Europol. Η Δανία είναι μια τρίτη χώρα σε αυτό το πλαίσιο και δεν θα μπορεί ε, να ασκήσει δικαιώματα ε, Λήψη αποφάσεων στα όργανα της Europol. Και βεβαίως ε, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι η Δανία θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σέγγεν, του χώρου Σέγγεν και η Δανία θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως την δανική νομοθεσία, την νομοθεσία, ε, την οδηγία περί δεδομένων και να δεχτεί επίσης την απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης και ε, την αρμοδιότητα ε, του, της Εποπτικής Αρχής ε, Προστασίας Δεδομένων. Όπως ξέρετε το Συμβούλιο, η Κομισιόν, η Δανία ξεκίνησαν μια νομική διαδικασία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια ομαλή διαδικασία, ίσως την 1η Μαΐου να είμαστε έτοιμοι. Ή έμπασε προς το συντομότερο δυνατόν μετά για να μπορέσουμε να ελεγχιστοποιήσουμε και να μηδενίσουμε ε, το όποιο κενό μπορεί να προκύψει από την 1η Μαΐου έως τη θέση σε ισχύ της μελλοντική Επικρισιακής Συμφωνίας. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Δανείοι εταίροι μας και αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος μεταφέροντας την νομοθεσία, την νέα νομοθεσία την προστασία δεδομένων που θα πρέπει να είναι έτοιμη στην 1η Μαΐου. Ο συνάδελφος από τη Δανία θα αναφερθεί σχετικά. Γνωρίζουμε ότι οι Δανείοι πολίτες θεωρούν ότι η συνεργασία με την Europol είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε για να βρεθεί μια λύση να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Το σχέδιο απόφασης ε, του Συμβουλίου ε, θέλει να προσθέσει τη Δανία στον κατάλογο των χωρών με τις οποίες μπορεί να υπάρξει ε, συμφωνία. Είναι το πρώτο βήμα αυτό. Θα θέλαμε να ακούσουμε βεβαίως τις ανησυχίες, τις επιθυμίες των μελών της Επιτροπής σας πολύ προσεκτικά και θα τα λάβουμε υπόψη μας αυτά όσο γίνεται νωρίτερα στη διαδικασία τη διαπραγματευτική. Οπότε ε, αναμένουμε τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε ε, στην Προεδρία του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη, αξιότιμα μέλη, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να δομήσω την παρέμβασή μου ω εξή. Πρώτα θα αναφερθώ στα βήματα που ακολουθήθηκαν μετά τη δήλωση της 15 η Δεκεμβρίου του 2016, την ίδια δηλαδή δήλωση στην οποία αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια θα σα δώσω κάποια στοιχεία που υπογραμμίζουν τη σημασία τη συνεισφορά τη Δανία στη Europol οπότε και την συνεισφορά για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και στη συνέχεια θα αναφερθώ στα βήματα που θα ακολουθηθούν μετά την σημαντική σημερινή ημέρα. Θα ήθελα να κρατήσω σαφές ότι έρχομαι εδώ με την πρόθεση να σας ακούσω και βεβαίως ε, ε, τα σχόλια και τις προτάσεις σας ε, να τα μεταφέρω Λοιπόν, τι έχει γίνει ως τώρα. Η διαδικασία ξεκινάει 15 Δεκεμβρίου 2016 με τη δήλωση. Στη δήλωση αυτή λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Δανία θα ξεκινήσουν τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν και θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες δράσεις μεταξύ των οποίων και επαφές με τους εμπλεκ, τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς. Στο άρθρο 26 της απόφασης της Europol, το σημείο φετηρίας στους, που αφορά τους κανόνες των σχέσεων της Europol προβλέπει ένα κατάλογο τον οποίο ε, εκπονεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν γρήγορα το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε την ε, εσωτερική διαδικασία και έστειλε μια επιστολή που ε, ζητάει τη συμπερίληψη της Δανίας ε, στο κατάλογο των τρίτων χωρών εστάλει από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο την 21η Δεκεμβρίου του 2016. Αμέσως μετά το Συμβούλιο μέσω ιστορικής διαδικασίας προετοίμασε μια εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου που έχει σταλεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 5 Ιανουαρίου Αξιότιμα μέλη, επιτρέψτε μου να σας δώσω παραδείγματα σε ό,τι αφορά την πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στη Δανία και την Europol. Το σύστημα πληροφοριών της Europol, γνωστό ως EIS, που είναι και βασική βάση δεδομένων της Europol, το 2016, το 2016 λοιπόν η Δανία ε, έκανε 19.000 αναζητήσεις στη βάση δεδομένων τέταρτη χώρα στην Ένωση ε, ανεξάρτητα το μέγεθος της χώρας. Επίσης έγινε αναφορά στα σημεία εστίασης. Όντως, η Δανία συμμετείχε σε 25 από τα 29 σημεία εστίασης στα focal points και συμμετέχει ενεργά. Σε ό,τι αφορά τη Σιένα τώρα, το σύστημα ανταλλαγή ε, ανταλλαγής μηνυμάτων, η Δανία το χρησιμοποιεί ενεργά. Το 2016 αντίλαξε πάνω από 15.000 μηνύματα αύξηση δηλαδή στάξεως του 11% σε σχέση με το 2015. Αυτή η αύξηση ε, ευθυγραμμίζεται και με τις ε, εκκλήσεις που έχουν γίνει ε, για την βελτίωση της λαγής πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα μέσω σχένα, η Δανία είναι ιδιαίτερα ενεργή στους τομείς της προτεραιότητας, τρομοκρατία, κλοπή και παράνομη μετανάστευση. Το 2016 η Δανία αντίλαξε 25% όλων των μηνυμάτων που έχουν να κάνουν με ληστείες. Στον τομέα της τρομοκρατίας αντίλαξε 15%. Για την παράνομη μετανάστευση 13% όλων των μηνυμάτων σχένα αφορούσαν και τη Δανία. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς εύκολα να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η Δανία όντως είναι μια χώρα που όντως μοιράζεται ε, στοιχεία με τη Europol. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην επιτρέψουμε επιχειρησιακά κενά από την 1η Μαΐου του 2017 και μετά. Και αυτό με οδηγεί στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της παρέμβασής μου. Θα ήθελα να, πω, να αναφερθώ στα μελλοντικά βήματα. Ξέρω ότι επήγει πολύ το θέμα. Εστάλει μια επιστολή ε, και στο Κοινοβούλιο ζητεί το Συμβούλιο από το Κοινοβούλιο τη γνώμη του το συντομότερο δυνατόν ή δυνατόν εντός ενός μήνα. Στη συνέχεια, όπως είπε πολύ σωστά και ο Πρόεδρος, θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο, δηλαδή στην ίδια τη συμφωνία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γυροπολ και θα υποβληθεί στο Συμβούλιο πριν το Συμβούλιο εγκρίνει την απόφαση αυτή και πάλι θα υπάρξει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το βήμα, η Europol και η Δανία θα μπορούν να συνάψουν και να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία ε, πριν από την 1η Μαΐου, ελπίζουμε. Έγινε ήδη αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σημασία του Πρωτοκόλου 22. Ο μόνος τρόπος η Δανία να συμμετάσχει πλήρως στον νέο κανονισμό Europol είναι να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο 22 των συνθήκων. Έτσι λοιπόν η Δανία δεν θα μπορεί να προσυμμετάσχει, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, όμως σε πλαίσια αυτής της μελλοντικής συμφωνίας θα επιτρέπει την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων έτσι ώστε να αποφύγουμε τα επιχειρησιακά κενά. Αξιότιμα μέλη, αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα, στην κατάληξη της ομιλίας μου. Χαίρομαι που σας παρουσιάζω εδώ το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και αναμένω περαιτέρω συνεργασία μαζί σας για αυτό το επίγον ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Δανικής Αρχής, στην εκπρόσωπο της Δανικής Αρχής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, θερμά την Επιτροπή σας που κάλεσε τις δανεικές αρχές να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση. Όπως ε, ανέφεραν και οι συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο η Δανία δεν μπορεί να συμμετάσχει στον κανονισμό της Europol από την 1η Μαΐου και μετά είναι το πρωτόκολλο 22 αυτό σημαίνει ότι η Δανία πλέον δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό της Europol και την εφαρμογή της. εφαρμογή του. Η λησαγωνοποίηση της Europol ήταν ένα από τους βασικούς λόγους ε, που οδήγησε στο δημοψήφισμα της, ε, του Δεκεμβρίου του 2015. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όμως ήταν αρνητικό είναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η δανική κυβέρνηση σέβεται πλήρως την απόφαση, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η δανική κυβέρνηση θεωρεί ότι το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα αυτό δεν απορρίπτει σε καμιά περίπτωση το σημαντικό έργο της Europol. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το το Δανικό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να φτάσουμε σε μια επιχειρησιακή συμφωνία με την Europol. Όλα τα κόμματα, ακόμα και αυτά που ήταν υπέρ του να περάσουμε από το opt-out σε opt-in, υποστηρίζουν ε, την δήλωση της 15 Δεκεμβρίου και τις λύσεις ε, που ε, έχει κατά νου. Είναι ένα ζήτημα κοινή ευθύνη αυτό. Η στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και αρχών υποβολής του νόμου, και υπηρεσιών ασφαλεία είναι κρίσιμη για τη συλλογική ασφάλεια τη Ένωση. Η Europol παίζει έναν, έναν κρίσιμο ρόλο, υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ε, και αρχών επιβολής του νόμου των χωρών αυτών. Η Δανία ήταν μέλο τη Europol από τότε που υπάρχει ε, η Europol και όλα αυτά τα χρόνια η Δανία συνεισφέρει πλήρως ε, και πιστά στη συνεργασία αυτή. Και βεβαίως η Δανία, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ε, παρέχει πολλά στοιχεία στο σύστημα πληροφοριών της Europol. Το 2014 και το 2015 ήμασταν από τα κράτη-μέλη που ε, διενέργησαν τις περισσότερες αναζητήσεις ε, στο EIS. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί η συνεργασία με την Europol και για τη Δανία και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ένωσης. Είναι προς συμφέρον όλων να εξασφαλίσουμε την συνέχιση της ταινής αυτής της συνεργασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αλλά και να προλάβουμε το δυσυνορικό έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία. Χωρίς μια επιχειρησιακή συμφωνία η Δανία θα γίνει ένας αδύναμος κρίκος στο σύστημα ασφαλείας της Ένωσης. Θα συμφωνήσετε όλοι ότι αυτό το σενάριο θα ήταν ατυχές ε, και μη επιθυμητό. Το αποτέλεσμα της ε, αποχώρησης της Δανίας από την Europol οδήγησε σε μια συζήτηση με την Κομισιόν για να βρούμε μια λύση. Συμφωνήσαμε με την Κομισιόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια επιχειρησιακή συμφωνία που να ελαχιστοποιεί τι αρνητικέ επιπτώσει ε, της τη δανεική αποχώρηση από την Europol. Αυτό ο επιχειρησιακό διακανονισμό ε, θα αφορά μόνο τη Δανία και βεβαίω δεν περιλαμβάνει πλήρη συμμετοχή στο Europol. Θα δημιουργήσει όμως ένα πλαίσιο για μελλοντική συνεργασία μεταξύ Δανίας και Europol. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Δανία θα εφαρμόσει την οδηγία για την προστασία δεδομένων πριν από την 1η Μαΐου του 2017. Θα υπάρξει απόφαση από αυτού, θα η οποία θα περάσει από το Κοινοβούλιο σύντομα. Η επιχειρησιακή συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έω την 1η Μαου όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέο κανονισμό Europol. Αυτό σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά σφιχτό. Βεβαίω αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρειαστείτε χρόνο και εσεί να αναλύσετε και να συζητήσετε το σχέδιο κειμένου. Η ιδανική κυβέρνηση θα σα βοηθήσει όσο μπορεί και είμαστε διαρρυθμένοι να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much to all three of... Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Έξι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Άλλος κανείς παρακαλώ. Έξι ομιλητές, δύο λεπτά ο καθένας, για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις των καλεσμένων μας και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και να κάνω και την ενημέρωση για την συνεδρίαση των συντονιστών. Ξεκινάμε με τον κύριο Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι μας κάνετε μια πολύ σωστή εξήγηση και διευκρίνηση της κατάστασης μας διευκρινίσατε και τα διαδικαστικά και τα ουσιαστικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά διαδικαστικά θέματα, η σύνεση και η μετριοπάθεια με υποχρεώνουν και μετριοφροσύνη με υποχρεώνουν να λάβω το λόγο γιατί ήμουν εισηγητής της ε, απόφασης του Συμβουλίου που καλύπτει ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο της Europol και επίσης ήμουν και ο εισηγητής για τον κανονισμό της ε, Europol που θα τεθεί σε ισχύ την 1η, 1η, την 1η Μαΐου συγγνώμη, 2017. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τις παρουσιάσεις και του Συμβουλίου και της Επιτροπής και της εκπροσώπου της ε, δανεικής κυβέρνησης και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι η Δανία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Επαναλαμβάνω, η Δανία είναι θεμελιώδης παράγον της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Επίσης, δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω καμία οικοτολογία. Ε, αλλά προβλέπω δύο οργανική συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων προτάθηκαν διάφορες ε, μορφές τέτοιες ε, απόφασης και φυσικά τρέφω από τον απόλυτο σεβασμό στην απόφαση της Λαϊκής Ιστανικής Ετοιμιγωρίας ε, του δημοψηφίσματος του, της 3ης Δεκεμβρίου και μάλιστα είχα την τύχη και το προνόμιο να μιλήσω εκτενώς με τον αξιοσέβαστο φίλο μου Μόρτεν Πέτερσον που όχι μόνο γνωρίζει κάλλιστα την Ευρωπόλ, αλλά είναι και πατριώτης ταυτόχρονα. Επίσης, συζήτησα δύο φορές με τον πρέσβη της Τανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την περασμένη εβδομάδα είχα την τιμή να μιλήσω και με τον Υπουργό Δικαιοσύνη σας. Οπότε είμαι απόλυτα εξοικειωμένο με την ουσία του θέματος. Πιστεύω ειλικρινά ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι σωστές και για τον τύπο και για την ουσία και η σπουδή είναι απαραίτητη γιατί θα χρειαστούν δύο ή τρεις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα πριν την 1η Πέμπτου, πριν την 1η Μαΐου. Οπότε ο χρόνος μας πιέζει για να μπορέσει η Δανία να εξακολουθήσει να διαδραματίζει το ρόλο της, το ρόλο ενός σημαντικού παράγοντα για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Μια ναι, και μας έδωσε δίλεπτο ο πρόεδρος, θα προσπαθήσω να το σεβαστώ. Πολύ καλή η διακήρυξη της 15ης Δεκεμβρίου, καλή η τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου, ώστε η Δανία ε, να είναι τρίτη χώρα χωρίς να είναι ουσιαστικά τρίτη χώρα. Εξομοιώνεται όμω με τρίτη χώρα και επίση ε, είναι καλή και συμφωνία επιχειρησιακή συνεργασία. Παρόλο που γνωρίζω τα όρια μια τέτοια επιχειρησιακή συμφωνία και φέρονται στη μη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα όρια. Δεν θα σας κουράσω με την απαρίθμηση αυτό το θέμα των ορίων. Πάντως χαιρετίζω αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι εμπρόθεσμα θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλους αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστούμε κύριε Διασταμέρα. Πολύ χρήσιμη η ενημέρωσή σας. Ο κύριος Πίτερσον. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη μετρική μου γλώσσα τα δανέζικα. Η Δανία χρειάζεται τη βοήθειά σας, γιατί αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Και ευελπιστώ ότι θα καταφέρατε, θα καταφέρετε να βοηθήσετε τη Δανία να αποχωρήσει πλήρως από τον κανονισμό της Europol, όπως θα γίνει από την 1η Πέμπτου του 2017. Και είναι δικό μας το σφάλμα. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιλογής που έγινε στο περσινό δημοψήφισμα τότε το δανεικό εκλογικό σώμα παραπλανήθηκε και νόμιζε ότι θα παραμείνει πλήρες μέλος ε, της Europol, κάτι που δεν ευσταθεί. Πάντω όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι προ το συμφέρον ούτε τη Δανία ούτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξωστρακιστεί πλήρω ε, από την Ευρωπόλη Δανία, γιατί συμβάλλει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματο και, και τη τρομοκρατία και η Δανία. Και έτσι με το σύστημα αυτό ε, θα είμαστε outsider τη Europol. Θα είμαστε μέλος ε, δεύτερη κατηγορία για την Europol, κάτι που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πάντω, σε αυτή τη φάση στηρίζω την διασύνδεση της Δανίας με τη Europol, παρόλο που δεν είναι ιδανική, δεν είναι τόσο καλό όσο ήταν και θα συνεχίσω τις προσπάθειές μας στο μέλλον η, Ευρω... Δανία να ξαναγίνει πλήρες μέλος της Ευρωπόλ, γιατί κάτι τέτοιο θα ωφελήσει και τους Δανούς πολίτες και τους υπόλοιπους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα, εμείς είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι, εμείς είμαστε υπέτοιοι για αυτή την κατάσταση και θα ήθελα επευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές για την κατανόηση που έδειξαν και την προθυμία τους ε, να επιλύσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία περίλθει η πατρίδα μου. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ καρποφόρα και επικοδομητική μας συνεργασία. Η κυρία Ζίπελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που τις περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι διασυνοριακό για να έχουμε τέτοια αποτελεσματική καταπολέμηση χρειαζόμαστε αποτελεσματική συνεργασία. Είναι αδύνατο να καταπολεμήσουμε το, το οργανωμένο έγκλημα μόνο με εθνικά μέτρα, με εθνικά τεκμήρια και χωρί συνεργασία. Η συνεργασία αυτή είναι απολύτω απαραίτητη. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα να επισημάνω και να ενισχύσω το επιχείρημα του κυρίου Μόρτεσεν. Το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Είναι ιδιαίτερα μείζον πολιτικό ζήτημα. Γιατί λοιπόν, αφού θέλουμε ε, να εμπλέξουμε τη Δανία, τα πολιτικά κόμματα και το, το δανεικό λαό, γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο θέμα να πάει σε δημοψήφισμα και στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτόμαστε πώ χειριζόμαστε τα δημοψηφίσματα. Γιατί τώρα βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε παρά το αποτέλεσμα του δημοψήφισμα, ε, το δημοψηφίσματος να βρούμε κάποια τεχνάσματα για να ξανακάνουμε τη Δανία τμήμα της Europol, αν και το δημοψήφισμα έλεγε να αποχωρήσει από αυτήν. Νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικό ζήτημα. Και έχουμε και ένα άλλο πολιτικό ζήτημα. Εγώ ανακαθεν πίστευα ότι όταν κανείς είναι μέλο μια λέσχη πρέπει να αποδέχεται του κανόνε που ισχύουν στη λέσχη αυτή. Κάτι που δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί επαριλημμένω είχαμε ρήτρε αυτοεξαίρεση opt-out. Λέει ένα, θέλω να είμαι σε αυτή τη λέσχη, αλλά θέλω για μένα να ισχύουν διαφορετικού κανόνε. Είναι δυνατόν σε λέσχε δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώ συγκροτούμε τη συνεργασία μα. Επίση, δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι η Δανία έγινε ξαφνικά τρίτη χώρα. Θα ήθελα να μας πει η νομική υπηρεσία πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, αυτή η εξομοίωση της Δανίας με τρίτη χώρα. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ασφάλεια δικαίου στα θέματα αυτά. Επίσης, ε, η σεπήρωση των οποίων είπε ο κύριος Πίτερσεν, ε, θεωρώ ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να ισχύει στο δυναικές. Συμφωνώ ότι σε κάποιο βαθμό θα πρέπει ε, η Δανία να είναι μέλος τη. Ευρωπόλ, όχι πλήρες μέλος όπως οι υπόλοιπες χώρες βέβαια, αλλά θα ήθελα να επιτευχθεί κάποια συμφωνία ή να γίνουν κάποιες δηλώσεις ή να υποβληθούν προτάσεις ώστε μακροπρόθεσμα να ξαναγίνει η Δανία πλήρες μέλος της Ευρωπόλ και να μην συνεχίσει την επόμενη 20 ετία να ισχύει ένα τέτοιο παράλογο ε, σύστημα με παρανοϊκές λύσεις σαν αυτές που προτείνονται τώρα. Ίσως να έχουμε μια ρήτρα σταδιακής εκπνοής ώστε κάποια στιγμή να γίνει και η Δανία πλήρες μέλος της Europol και να αποφύγουμε αυτά τα περίεργα τεχνάσματα που επινοούμε τώρα. Θα ήθελα να πω κάτι και για τους συντονίστες μετά. Η κυρία Έρνστ. Σας ευχαριστώ. Δύσκολο όντως το θέμα ακαθόδες και θα οφείλουμε να σεβαστούμε το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Τώρα, πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση θα το δούμε. Πάντως, η συζήτηση είναι απόλυτα εύλογη και θεμητή, παρόλο που δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί είναι δύσκολο να υποβάλουμε σε δημοψήφισμα τόσο περίπλοκες συμφωνίες. Αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Ε, είναι εθνικό ζήτημα για το τι ερωτήματα θα μπαίνουν και τι ζητήματα θα μπαίνουν σε δημοψήφισμα. Στην ε, ομάδα μας δεν είμαστε και πολύ ενθουσιώδεις απέναντι στην ε, Europol. Έχουμε επικρίσεις και προβλήματα και με τη διεξαγωγή των ελέγχων, αλλά είναι λογικό η προσπάθεια καταπολέμησης ε, να γίνεται σε διασυνοριακό επίπεδο και με συνεργασία. Αυτό είναι πασιφανές ότι χρειάζεται. Τώρα, πώς θα εξέλθουμε από αυτό το αδιέξοδο. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Τι χαρακτηριστικά θα έχει η συμφωνία. Η Δανία δεν θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων αλλά θα συνεχίζεται η ανταλλαγή δεδομένων. Έχουμε και τις ε, συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων. Πώς θα ισχύσουν αυτές. Και η Δανία θα είναι μεν μέσα, αλλά θα εξομοιώνεται με τρίτη χώρα. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω όλα αυτά. Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Και επίσης να γίνει μια εμπεριστατωμένη και ενδελεχής ανάλυση των προτάσεων. Ελπίζω πόντως ε, να τα καταφέρουμε και να προλάβουμε πριν την 1η Μαΐου να ετοιμαστούμε. Εξετάζονται διάφορα σενάρια και σίγουρα είναι συμφέρον μας να βρούμε λύση. Και έχουμε και μια, ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δανικού Κοινοβουλίου που ζητά σύναψη κάποιε συμφωνίες με την Ευρωπόλ, δεν πρόκειται να τον μπλοκάρουμε, αλλά υπάρχει και μια φαιά σε όλα αυτά, μια σάφια. Μήπως ε, τελικά οδεύουμε προς μια ε, εξέλιξη που είναι απευκταία, που είναι οι διαφορετικέ ταχύτητε και η μεγάλη διαφοροποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θέλουμε διευκρινήσει και κάποιε νομικέ αποσαφηνήσει. Ο κύριος ECR-gruppen har altid respekteret øh, princippet omkring... Ευχαριστώ. Η ομάδα ECR ήταν ανέκαθεν υπέρ της ιδέας της ε, αυτοδιάθεσης, αυτοπροσδιορισμού και του δικαιώματος ε, των λαών να επιλέξουν την πορεία και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχουμε και τι ρήτρε αυτοεξαίρεση. Έχουμε τη Βρετανική ρήτρα αυτοεξαίρεση, τη Δανική, αλλά και άλλε χώρε έχουν αυτοεξαιρέσει για επιμέρου τομεί. Θέλουμε μία κατάσταση όπου συμφωνία μεταξύ Δανική κυβέρνηση και Συμβουλίου και Επιτροπής να, να ήταν ευρύτερη. Βέβαια, συμφωνούμε γιατί στη Δανική Βουλή υπάρχει διακομματική συμφωνία υπέρ της εφαρμογής της ε, συμφωνίας αυτής Δανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκ μέρους της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θα στηρίξω αυτή τη διαδικασία, θα την υπερψηφίσω και ελπίζω να έχουμε ομαλές εξελίξεις και το συντομότερο δυνατό, αφού γίνει η αποσαφήνιση των νομικών θεμάτων. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία εμπρόθεσμα, πριν δηλαδή την κέρια αυτή διορία της 1ης Μαΐου του 2017. Εμείς θα συμβάλλουμε στην προώθηση αυτού του θέματος. Και ο κύριος, ε, ο κύριος Μπέγκστον, παρακαλώ. Thank you, Chair. I will also speak in uh, my mother tongue. Θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κόμματα εκείνα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα η Δανία να συνεχίσει να επιχειρεί εντό τη Europol. Όμω, όπω συνάδελφο ο κ. Πίτερσεν, πρέπει να πω ότι θα είναι έτσι μια συμμετοχή δεύτερη κατηγορία. Θα είμαστε μέλο δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Δεν θα έχουμε άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων, ε, ούτε στις επιχειρήσεις ε, και ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ίσως να μην έχει και πολύ νόημα ε, σε, για πολλούς από εμά αυτό. Δεν θα είμαστε λοιπόν πλήρες μέλος της Europol. Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ελπίζω να γίνει κάποιο άλλο δημοψήφισμα κάποια άλλη στιγμή για να ξαναγίνουμε πλήρες μέλος της Europol. Μάλιστα. Νομίζω οι συνεισφορές σας ε, ήταν αρκετά σαφείς Δεν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες νομίζω. Ο καθένας εξέφρασε τις θέσεις του. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να απαντήσει σε κάτι. Λουίτζι πρώτα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη που πήραν το λόγο διότι η φωνή των ανησυχιών σας είναι σημαντική για μας εμείς θα υποστηρίξουμε την Europol για να συμμετάσχει στην επικοινωνιακή συμφωνία και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα αυτά που πρέπει για την προστασία δεδομένων. Και ακούγοντας ε, την επιβεβαίωση ε, από τη δανεική κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστεί η νομοθεσία που προστασίας δεδομένων, από την νομοθεσία πριν την 1η Μαΐου, ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και μας καθυσυχάζει. Η κυρία Σίπελ τώρα ανέφερε κάτι σημαντικό, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας. Η ανησυχία σχετικά με τον περιορισμένο χρόνο ε, της υπηρεσιακής συνεργασίας. Ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι ε, πόσο σημαντική είναι η Δανία ως εταίρος μας στα ζητήματα ασφαλείας και πόσο σημαντικό θα είναι πιο μακροπρόθεσμα να δούμε πώς η Δανία μπορεί να βελτιώσει τη συνεργασία της με την Europol. Θα πρέπει λοιπόν να, θα πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριλάβουμε μια ρήτρα αναθεώρηση στη συμφωνία, να υπάρξει κάποια έκθεση αξιολόγηση για να δούμε πώς θα προχωρήσει η εφαρμογή αυτής της υπηρεσιακής ε, συμφωνίας. Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε η Δανία να συμμετάσχει πλήρως ε, στο νέο κανονισμό Europol είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο 22. Υπάρχει βεβαίως περιθώριο βελτίωσης, εμείς είμαστε ανοιχτοί ε, για να συμβεί αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχει το πρωτόκολλο 22, υπάρχουν οι κανόνες ε, οι οποίοι και εφαρμόζονται πλήρως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μάλιστα δεν ξέρω αν θέλουν να απαντήσουν οι ιδανικέ αρχέ, η Προεδρία. Η Προεδρία. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δίας Δεμέρα για αυτά που είπε. Ε, πραγματικά ήταν ε, μια παρέμβαση ε, υπεύθυνου πολιτικού παράγοντα. Απαντήθηκε αυτά που είπε η κυρία Σίπερ από την Επικόσπο τη Κομισιόν για την προστασία δεδομένων αν εξτάσει κανείς τη δήλωση, και στην πρώτη παράγραφο λέγεται ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο επικοινωνιακής συνεργασίας των οποίων που θα περιλαμβάνει μεταξύ των οποίων και ανταλλαγή δεδομένων με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Εφόσον αποτυπώνεται λοιπόν το πνεύμα αυτής της ε, δήλωσης ε, στη συμφωνία, νομίζω ε, δεν έχουμε λόγο ανησυχίας. Μάλιστα, να ευχαριστήσω τους τρεις προσκεκλημένους. Ε, θέλω να, διασφαλίσω στους συναδέλφους ότι η προσέγγιση ε, ήταν εξαιρετικά προσεκτική κατά την προπαρασκευή της συνάντησης. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, δεν θα σχολιάσω εγώ την πολιτική κατάσταση που μας έφερε ως εδώ, αλλά η θέση είναι η εξής. Τα πιο έμπειρα μέλη το είπαν σαφέστατα και ο προηγούμενος συζητητής ε, για την Europol. Οι συντονιστές τώρα θα πρέπει να ορίσουν έναν εισηγητή για την γνωμοδότηση. Ο κύριος Διαδεμέρα αλλά και άλλοι αναφέρθηκαν στην νομική πτυχή μίλησαν είπαν ότι πρέπει να όλοι να επιδείξουμε αίσθημα ευθύνης, να κινηθούμε γρήγορα. Βεβαίως είναι μια απόφαση που μπορούν να πάρουν οι συντονιστές σήμερα. Αυτό που έχει σημασία αγαπητοί συνάδελφοι είναι να υπάρξουν δεσμεύσεις από τη Δανία. και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, τη μεταφορά της οδηγίας ε, για τη, σημαντική, για τη συμμετοχή στη Σέγγεν υπάρχει και η εφαρμογή της νομολογίας του δικαστηρίου για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρησιακές ε, ε, ανάγκες αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Europol και Δανίας για λόγους ασφάλειας πολλές συναντήσεις έχουν γίνει από αυτού αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι είναι θέμα σημαντικό αλλά πρέπει να είμαστε και σαφείς η πρόταση αυτή ουσιαστικά αφαιρεί αρμοδιότητες από το Κοινοβούλιο για ένα ζήτημα που αφορά τον τρίτο πυλώνα πρώτης Λισαβόνας. Αυτό αποτελεί εξαίρεση. Ε, το είπαν εδώ σήμερα και τα πιο έμπειρα μέλη. Η λύση λοιπόν που θα βρεθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να μετατρέψει αυτές τις εφαρμοστικές αποφάσεις του Συμβουλίου σε ένα νομικό μέσο που να ευθυγραμμίζεται με τον νέο κανονισμό. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να πάμε προς κάτι καλύτερο από νομικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση, επίγουσα, θα κάνουμε το καθήκον μας, θα ορίσουμε έναν εισηγητή ε, μετά από τις συστάσεις και των συντονιστών σήμερα το απόγευμα στα πλαίσια αυτά τα χρονικά, τα σφιχτά που έχουμε. Θα το συζητήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την ε, τοποθέτηση τους την εξαιρετικά μετρημένη και το, το ότι έχουν αντιληφθεί την εξαιρετική κατάσταση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Μετά τις συναντήσει με τους συντονιστές θα σας ενημερώσω για τις εξελίξεις.